Λοιπόν. Ο κύριος Περχόφστερ. Η συζήτηση αυτή αφορά το τι μπορούμε να περιμένουμε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Πέμπτης και της Παρασκευής. Οπότε αυτό το οποίο ελπίζω εγώ και η ομάδα μου και η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου αυτού είναι να τελειώσει αυτή η σύνοδος κορυφής, κύριε Μπαρόζο, με πιο αποφασιστική και τολμηρή προσέγγιση στην ε, κρίση αυτή. Γιατί, ας είμαστε αυτή τη στιγμή συνολική αντιμετώπιση της κρίσης δεν υπάρχει. Ούτε από πλευρά Συμβουλίου, ούτε από πλευρά ε, Κοινοβουλίου. Και Ανέφερε κάποια ερωτήματα ο κύριος Σούλτ για τους οίκους και το ρόλο τους στην κρίση αυτή. Αλλά ας προσπαθήσουμε να βρούμε τις πηγές της κρίσης και τα σφάλματα, όπως λέει και ο Σέξπιρ, στον εαυτό μας. Εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η κρίση δεν έχει τελειώσει. Όσοι θεωρούν πως με το να δώσουμε περισσότερα χρήματα στην Ελλάδα θα ε, τελειώσει η κρίση της Ελλάδας και του ευρώ, έχουν λάθος. Η κρίση δεν έχει τελειώσει. Η κρίση θα συνεχιστεί εάν πρώτα απ' όλα δεν βρούμε μια δομική διαρθρωτική λύση για την ε, Ελλάδα και δεύτερον εάν δεν δημιουργήσουμε πραγματική Ευρωπαϊκή και Οικονομική Ένωση στην Ευρώπη. Έτσι θα τελειώσει η κρίση του ευρώ και τη Ελλάδα. Γιατί, και πάλι, είναι δυνατόν να έχουμε ένα νόμισμα και 17 κυβερνήσει, 17 οικονομικέ στρατηγικέ, 17 αγορέ ομολόγων. Αυτό δεν γίνεται πουθενά στον κόσμο. Μόνο εμείς στην Ευρώπη νομίζουμε πώς μπορούμε να έχουμε νομισματική ένωση και 17 διαφορετικές κυβερνήσεις, πολιτικές και αγορές ομολόγων. Και μόνο εμείς ως ε, φεντεραλιστές το λέγαμε εμείς αυτό. Χτες ο κύριος Λίψκι, διευθύνων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ζήτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση να δημιουργήσει πολιτική και οικονομική ένωση. Χτες ο κύριος Γκάιτνερ, Υπουργός Οικονομικών, τον είπα, που είπε ίσως ε, να συζητήσουν και να δημιουργήσουν μια πολιτική και οικονομική ένωση. Εάν στην άλλη όχθη του Ατλαντικού ξέρουν τι πρέπει να κάνουμε, εμείς γιατί δεν έχουμε το θάρρος να κάνουμε αυτό το τεράστιο βήμα προς τα μπρος για μια οικονομική και πολιτική ένωση, κύριε Πρόεδρε. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα για το Αυριανό Συμβούλιο. Και θεωρώ, και αυτό είναι το δεύτερον, πρέπει να βοηθήσουμε την Ελλάδα, όχι μόνο αμυντικά, να υπάρξει ένα τολμηρό πρόγραμμα λιτότητας, αυτό το οποίο συζητιέται αυτή τη στιγμή με την ελληνική κυβέρνηση και ίσως υπάρχουν ιδέες για να πάμε ακόμη παραπέρα από αυτά τα οποία υπάρχουν επιτάπτως, αλλά πρέπει να υπάρχει και ένα θετικό σχέδιο. Δεν μπορούν να βγουν από την κρίση μόνο με τη λιτότητα. Χρειάζεται ανάπτυξη και επενδύσεις. Και αυτό μπορεί να γίνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Α δώσουμε παραδείγματο χάρη εγγυήσει για ιδιωτικέ επενδύσει. Δεν υπάρχουν πια ιδιωτικέ επενδύσει στην Ελλάδα. Επίσης δάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Και γιατί να μην χρησιμοποιήσουμε μέρος των ιδιωτικοποιήσεων όχι μόνο για την εξυγίανση του προϋπολογισμού, αλλά για νέες επενδύσεις και ανάπτυξη στην Ελλάδα. Έχω ε, ένα αίτημα ε, και μία ερώτηση όχι για τον κύριο Σούλτ αλλά και τον κύριο Ντόλ. Θα τα πω γαλλικά. Θα πρέπει να είμαστε πολύ σαφείς επί του θέματος. Εάν θέλουμε να δώσουμε χρήματα στην Ελλάδα, θα πρέπει να υπάρξει πολιτική συνένεση στην Ελλάδα για να δώσουν οι υπόλοιπε χώρε ε, χρήματα. Και θα ήθελα να κάνω έκκληση στον κύριο Ντόλ που είπε πράγματα τα οποία ήταν λυθή να πείσει του πολιτικού του φίλου να δώσουν αυτή την πολιτική συνένεση για να υπάρξει ε, συνέχεια για την Ελλάδα. Το χρειαζόμαστε αυτό. Το ξέρω ότι είναι πολύ βαρύ το καθήκον που σας αναθέτουμε, Ζόζεφ, αλλά νομίζω ότι είστε στο ύψος των ε, περιστάσεων και μπορείτε να το κάνετε, διότι πράγματι είναι αλήθεια η χώρα που βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση θα πρέπει να εμπνέει πολιτική ενότητα και δεν θα πρέπει να κάνουμε πολιτικά παιχνίδια σαν αυτά που γίνονται στην Ελλάδα. Και έχω την εμπειρία ως Βέλγος, ε, κύριε Λάγκε. Το γνωρίζω αυτό ως Βέλγος. Και τέλος, κύριε Πρόεδρε, Ας είμαστε και ειλικρινείς. Χρειάζεται ένα άλλο πακέτο οικονομικής ε, διακυβέρνησης από αυτό το οποίο προτείνουμε σήμερα. Και πρέπει να ρωτήσω κάτι ευθέω τον κύριο Μπαρόζο. Χτες ο εκπρόσωπο της Κομισιόν στην ε, συνέντευξη τύπου είπε πως δεν υπάρχει ανάγκη για αντίστροφη ειδική πλειοψηφία στο πακέτο διακυβέρνηση. Σας ζητώ να το διορθώσετε κύριε Μπαρόσο και ζητώ η Κομισιόν μαζί με το Κοινοβούλιο να ταχθεί υπέρ μιας πιο κοινοτική μεθόδου στο πακέτο οικονομικής διακυβέρνησης. Ευχαριστούμε κύριε Βερχώστα. Ε, θέσατε μια ερώτηση προς τον κύριο Ντόρ, ο οποίος θα ήθελε να ανταπαντήσει. Ε, ανακοίνησε, τη, την μπλε του κάρτα και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν δέχεστε να σας υποβάλει την ερώτηση ε, ο κύριος Ντόλ. Και επίσης έχει ζητήσει να σας ε, θέσει μια ερώτηση και ο κύριος Κουμουτσάκος. Συμφωνείτε? Ο κύριος Ντόλ πρώτα. Ναι βεβαίως και πολύ γρήγορα. Θα ήθελα να διατυπώσω εντάχει το ερώτημα προς τον πρόεδρο των φιλελευθέρων, της ομάδας των φιλελευθέρων. Τη μέρα που θα αναλάβει το παιχνίδι της αλληλεγγύης ονόματι των φιλελεύθερων κυβερνήσεων για όλες τις χώρες σας διαβεβαιώ ότι εγώ θα κερδίσω στον αγώνα αυτό εκ μέρους της ομάδας μου και στην Ελλάδα και θα είσαι εδώ και θα είμαι εδώ και θα τα ξαναπούμε. Κύριε Φερχόφστα, μπορείτε να απαντήσετε. Ναι, Πρόεδρε. Μια και στι περισσότερε χώρε, στι οποίε αναφέρεται ο κύριο Ντόλ, συμμετέχουμε σε κυβερνητικού συνασπισμού με του χριστιανοδημοκράτε. Ε, κάπου βοηθάμε κι εμεί από ό,τι φαίνεται. Εν πάση περιπτώσει όμως ε, τώρα το απόγευμα και πριν από ένα τόσο σημαντικό συμβούλιο δεν νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε ε, κουβέντα για κόμματα και να φέρνουμε τη μία κυβέρνηση απέναντι στην άλλη. Ζωζεφ, το θέμα δεν είναι να με φιλελεύθερη κατά του ΕΛΚ, κατά των σοσιαλιστών. Εγώ σου ζητώ, Ζωζεφ, να πείσει τους φίλους σου της Νέας Δημοκρατίας εκ των οποίων πολλούς γνωρίζω και εγώ προσωπικώς και έχουμε και κάποιους που ήρθαν στην ομάδα μας, θα ξέρεις, κάποιους. Λοιπόν, ένα πράγμα να κάνουν, ενότητα, συνένεση για να βγει ο λαός από την κρίση. Και έχεις και εσύ ρόλο να διαδραματίσεις αυτό. Στηρίζομαι στη συνεργασία σου. Ευχαριστώ το λόγο για κύριο Σκουμουτσάκος για ένα αίτημα ακόμη. Κύριε Βερχόφστατ. Θα σας παρακαλέσω μόνο σε 30 δευτερόλεπτα να δώσετε την απάντηση σας, κύριε Κουμουτσάκο. Χαρά άκουσα τον κύριο Πρόεδρο ότι όλοι πλέον έχουν, αντι... έχουν αντιληφθεί ότι το πρόβλημα της ελλάδας είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα. ποιο είναι το καθήκον της ελλάδας κύριε πρόεδρε; το καθήκον είναι να προχωρήσει τις διαρθρωτικές μεγάλες μεταρρυθμίσεις και να προχωρήσει σε ιδιωτικοποίησεις. θέλω λοιπόν να ενημερώσω τον κύριο πρόεδρο γιατί προφανώς είναι παραπληροφορημένος ότι στα δύο αυτά θέματα που είναι ο σκληρός πυρήνας των μεταρρυθμίσεων η νέα δημοκρατία όχι μόνο έχει συμφωνήσει είναι δικές της προτάσεις δικές της προτάσεις που η κυβέρνηση ενάμιση χρόνο τώρα αδυνατεί να πραγματοποιήσει. αυτή είναι η αλήθεια. Δεν είχατε ερώτηση κύριε Κουμουτσάκο, δήλωση ήταν αυτό μόνο. Ωραία λοιπόν. Κάνουμε ότι δεν ακούσαμε και δίνουμε το λόγο στο... στην κυρία... Στον κύριο, Ράντφορτ είναι μια ερώτηση. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ελπίζω να μ' ακούτε όλοι. Άκουσα με μεγάλη προσοχή τα λόγια του κύριου Φερχόφστατ. Κύριε Πρόεδρε. Και θα ήθελα να ρωτήσω εάν όντως το σύνθημά σα είναι ότι η Ελλάδα βρίσκεται παντού. Ότι δεν είναι ένα μεμονωμένο μόνο κράτο μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αποτελεί έκφραση ενό γενικότερου κλίματο, μια γενικότερη ατμόσφαιρα. Δηλαδή ότι η Ελλάδα είναι πανταχού. Κύριο Φερχόφιστα, απάντηση. Κύριε Πρόεδρε, θεωρώ πως είναι προφανές πως αν δεν λύσουμε το ελληνικό πρόβλημα θα έχουμε τεράστια προβλήματα σε ολόκληρη την Ευρωζώνη. Ήδη στην Πορτογαλία έχουμε, ήδη στην Ιρλανδία έχουμε. Ξέρετε πως η διαφορά στην ψαλίδα των ε, επιτοκίων είναι πάνω από 800 μονάδες βάσης μεταξύ Πορτογαλίας και Γερμανίας, Ιρλανδίας και Γερμανίας. Οπότε τι κάνουμε η αλληλεγγύη που χρειαζόμασταν στην αρχή της κρίσης και δεν υπήρχε, δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, πρέπει να είναι για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης. Και λόγω της έλλειψης αλληλεγγύης το Δεκέμβριο του 2009 δημιουργήσαμε πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα από το πρόβλημα αυτό που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Ευχαριστώ. Προχωράμε τώρα με τη συζήτηση. Ο λόγος στον κύριο Τιλ για δυόμιση λεπτά. Uh, thank you, Mr. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ διασκεδαστική ημέρα σήμερα εδώ στο Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να σας ε, υπενθυμίσω ότι πολλοί ημών έχουμε βιώσει κομμουνισμό. Και φαίνεται ότι έχουμε κάνει μια τεράστια και γρήγορη πρόοδο για να προετοιμαστούμε για την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειάστηκε να αποδείξουμε ότι μπορούμε να πληρώνουμε τα κριτήρια της Κοπενχάγης και μπορούμε να έχουμε πλήρως λειτουργούσες οικονομίες αγοράς και μία σειρά από άλλα κριτήρια. Δυστυχώς όμως αυτό ο, το επίπεδο ελέγχου δεν επευλήθη σε κάποια κράτη-μέλη όταν εντάχθηκαν στην Ευρωζώνη. Και γιατί αυτό? Γιατί δημιουργήθηκε ως πολιτικό και όχι ως οικονομικό πρόγραμμα. Επομένως αγνοήθηκαν κριτήρια, άλλαξαν στατιστικά στοιχεία για να ενταχθούν χώρες που δεν ήταν ακόμα έτοιμες και αυτό είναι και η ουσία του προβλήματος. Και αυτή τη στιγμή ζούμε τις συνέπειες και βρισκόμαστε και σε μια πολύ κρίσιμη καμπή. Παρά το γεγονός ότι τα περισσότερα μέλη της πολιτικής μου ομάδας είναι από χώρε μη μέλη της Ευρωζώνης, δεν θέλουμε να αποτύχει το ευρώ. Επίσης, δεν θεωρώ όμως ότι θα πρέπει να υπερασπιζόμαστε το ευρώ με κάθε τίμημα. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο λοιπόν αυτή τη φορά θα πρέπει να αποστείλει ένα σαφές μήνυμα και το μήνυμα είναι ότι αν κάποιος δεν μπορεί να σταθεί εντός της Ευρωζώνης τότε εάν δεν κάνει πολύ σημαντικές αλλαγές η Ευρωζώνη δεν θα πρέπει να διστάσει να θέσει ζήτημα αναδιάρθρωσης του χρέους τους ή όσο επάναυσο και αν ακούγεται να τον εκδιώξει από την κλειστή αυτή λέσχη. Εάν δεν το κάνετε αυτό, κύριε Πρόεδρε, να θα σας πω τι θα γίνει στη συνέχεια. Την επόμενη φορά, οι αντίπαλοι σας ή οι αντίπαλοι του διαδόχου σας δεν θα είναι καλοί και αξιοπρεπείς ευρωσκεπτικιστές όπως είμαι εγώ, αλλά αντιευρωπαίοι και μάλιστα κακοί αντιευρωπαίοι. Διότι θα έχουν εκλεγεί από ε, οργισμένους Γερμανούς φορολογούμενους, από ε, Ολλανδούς ε, ιδιωτικούς επιχειρηματίες που δεν θα αντέχουν άλλο να πληρώνουν τα χρέη των άλλων. Και ξέρω κύριε Πρόεδρε ότι αυτό δεν θέλετε να συμβεί ούτε εσείς ούτε εγώ. Ας δράσουμε όμως βάσει αυτού. Και κύριε Πρόεδρε θα ήθελα επίσης να σας ζητήσω να σταματήσετε να ε, κάνετε κατάχρηση κάθε κρίση προκειμένου να πείσετε να υπάρχει ακόμα περισσότερο υπερεθνικό πρόγραμμα, φορολογική ένωση και ούτω καθεξής, γιατί αυτά δεν μας βοηθούν. Δεν είναι κρίση της Ευρώπης αυτό, είναι κρίση μιας λανθασμένης, παροχημένης έννοιας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Και μόνον αυτό. Ευχαριστώ κύριε Ζαχράτηλ. Η κυρία Χάρμς έχει το λόγο. Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, αξιότιμη κυρία Γκέρι, αξιότιμοι συνάδελφοι. αισθάνομαι κατάπληξη για το πόσο ξαφνικά ε, συγκινητική γίνεται αυτή η συζήτηση για τη βαθύτατη κρίση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Νομισματικής Ένωσης που κρυβόταν τόσο καιρό και δεν τη βλέπαμε. όταν δεν μπορέσαμε εν ώψη της ανάληψης προεδρίας της Ουγγαρίας να λύσουμε το θέμα της ε, ελευθερίας του τύπου, όταν δεν μπορέσαμε εν ώψη της μεγάλης κρίσης στη Λιβύη και στα άλλα κράτη της περιοχής να εκφραστούμε με μία ενιαία φωνή, τι μπορούμε άλλο να κάνουμε στην περίπτωση της μεγάλης κρίσης που αντιμετωπίζει η Ελλάδα παρά να διαπιστώσουμε ότι ξαφνικά η Ευρώπη έχει πολλούς προέδρους αλλά κανέναν ηγέτη. Δεν έχει ηγεσία. Και αυτό είναι το πρόβλημα που πρέπει να συζητήσουμε και να αντιμετωπίσουμε. Γιατί μπαίνουμε όλο και πιο πολύ σε μια κρίση που διαρκεί περισσότερο από την ελληνική κρίση και το Συμβούλιο δεν δίνει απαντήσεις ή δεν τις δίνει εγκαίρως ή δεν τις δίνει στο επίπεδο των περιστάσεων. Το να μιλούμε μόνο για διάσωση της Ελλάδας ή μόνο για σταθεροποίηση του Νότου μπορεί να αποτελέσει τη μοναδική λύση για την Ευρώπη. Και ότι αρκεί για, την καλύτερη, για ένα καλύτερο επίπεδο διαβίωσης και για την ευημερία των Ευρωπαίων δεν έχει δοθεί σαν απάντηση. Υπάρχει ένα αρμόδιο όργανο το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Κοινοβούλιο έχει, θα έλεγα, μόνο κάποιες λαμπρές στιγμές, αλλά δεν ετόλμησε εγκαίρως πριν από το ιστορικό αυτό Συμβούλιο να συνέλθει για να διατυπώσει ψήφισμα μέσα στο οποίο θα περιέγραφε ακριβώς τα προβλήματα που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν εν αυτής της ιστορικής κρίσεως και λυπούμε ιδιαίτερος, ειδικά για τους συναδέλφους που βρίσκονται στα δεξιά μου και στα αριστερά έδρανα του Κοινοβουλίου, διότι δεν θέλησαν εγκαίρως να βοηθήσουν να δοθούν ουσιαστικές απαντήσεις απαντήσει από πλευρά του Κοινοβουλίου για την περίπτωση τη Ελλάδα. Θα ήθελα επίση να αναφερθώ και στα όσα είπατε εσεί για την περίπτωση τη Ελλάδα, Ο Γιώζεφ Ντάουλ έχει ευθύνη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, ναι. Αλλά για να είμαστε και δίκαιοι θα πρέπει να πούμε ότι και η σοσιαλιστική ομάδα αισθάνεται ότι έχει ευθύνη ενάντια του Παπανδρέου και τη κυβέρνησή του. Χαίρομαι που πήρε την ε, ψήφο εμπιστοσύνη εχθέ. Αλλά τα δίκαια προγράμματα, τα σωστά προγράμματα μέσα στην κρίση τα αποφασίζει η ελληνική κυβέρνηση. Τις αδικίες και την μετακύληση του δανείου, την φοροδιαφυγή, την ανεπαρκή διαχείριση των δημόσιων οικονομικών πάλι η Ελλάδα τη διαχειρίζεται και γι' αυτό θα πρέπει να μιλήσουμε ξεκάθαρα για τις διάφορες ελίτ στην Ελλάδα οι οποίες έχουν μεγάλο μερίδιο της ευθύνη για αυτή την βαθύτατη κρίση. Και υπόθηκε πολύ συχνά ότι χρειάζεται να υπάρχει μεγαλύτερο διάστημα αποπληρωμής του δαμηνίου, πιο ευνοϊκές συνθήκες, δηλαδή μία αναδιάταξη του δανείου, ήπια έστω, διακριτική μεν, αλλά για αυτήν δεν υπάρχει καν επαρκής πολιτική καθοδήγηση και ηγεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε αυτό το οποίο αναγνωρίστηκε εγκαίρως ως πρόβλημα, δηλαδή ως λύση, μάλλον ως συμμετοχή των ιδιωτών ε, δανειστών στην ε, ε, διαχείριση, στο δάνειο και που αποτέλεσε και την πηγή της κρίσης, διότι αυτό οδήγησε στην βάθηση της κρίσης, δεν το λέει κανείς. Και τώρα προβλέπετε πάλι προτείνεται πάλι σαν λύση και σαν διάσωση η συμμετοχή των ιδιωτών. Γι' αυτό λοιπόν κύριε Μπαρόζο, σας εύχομαι κάθε επιτυχία όταν λέτε ότι θα πρέπει να υπάρξει μια πιο δίκαιη φορολόγηση ως διέξοδος για την κρίση. Δεν ξέρω αν θα ακολουθήσετε την λύση της ε, φορολόγησης των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Εμείς ως ομάδα πάντοτε ήμασταν υπέρ ε, εδώ μέσα στο Κοινοβούλιο, αλλά η φοροδιαφυγή ή τα μεγάλα πριν που δίνονται στους, ε, στα στελέχη των επιχειρήσεων είναι σε μεγάλο βαθμό και, και αυτά ένα μέρος του προβλήματος και είναι και δική σας ευθύνη. Ευχαριστώ πολύ. Την κυρία Χάμψο, ο κύριος Μπίσκη, δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εάν δει κανεί στην Ελλάδα αυτές τις μέρες μπορεί να μάθει και κάτι. Με διαταγές ε, περί λιτότητας και με πληστηριασμό και των τελευταίων ασημικών του κράτους δεν σώζεται η Ελλάδα. Ε, τι να σου πω, αναλάβετε εσείς την ευθύνη τότε. Αλλά συνεχίζουν τα πράγματα ως έχουν. Πριν υποσχεθούμε οτιδήποτε, ζητάμε ακόμη περισσότερη λιτότητα και ιδιωτικοποίηση. Και είχαμε και αυτό το ευρωπαϊκό εξάμεινο το οποίο φαίνεται πως θα περάσει για τα κρατημέλη. Πάει δε τόσο πολύ μακριά η υπόθεση ώστε μιλάμε για σύσταση υπηρεσίας ιδιωτικοποιήσεων με πρότυπο το γερμανικό Τρόιχαντ που έκανε κάποια θετικά πράγματα αλλά οδήγησε και σε φοβερή αποβιομηχάνηση και ξέρετε πως ακόμα μέχρι σήμερα υπάρχουν τα σημάδια εκεί πέρα. Εγώ δεν θα είμαι τόσο αλαζόνας. Επιπλέον, περισσότερα δισεκατομμύρια για την Ελλάδα χωρίς να αλλάξει η πορεία είναι μόνο προστασία για τις τράπεζες. Επιπλέον, ακούσαμε πως δεν θα ζητηθεί ε, εθελοντική συμμετοχή των τραπεζών. Πλέον μιλάμε για πολιτικό ναυάγιο. Οπότε η μοναδική εναλλακτική για εμάς είναι ριζική αλλαγή στην οικονομική και χρηματοοικονομική πολιτική, αλλά λείπει το θάρρος γι' αυτό. Η αιτία της κρίσης δεν καταπολεμάται και αυτό είναι το πρόβλημά μας. Λείπει το θάρρος για περισσότερη δημοκρατία και διαφάνεια και λιγότερη πολιτική πίσω από κλειστέ πόρτες. Έτσι κινδυνεύει το ευρωπαϊκό ιδεώδες οι εθνικισμοί κερδίζουν έδαφος οπότε θα πρέπει από τις συνόδους κορυφής να στέλνονται ξεκάθαρα μηνύματα. Όχι το μήνυμα συνεχίζουμε όπως τώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Για δύο λεπτά ο κύριος Φάρατς Κύριε Πρόεδρε, κάθε φορά που σας ζητάω ποιο είναι το εναλλακτικό σας σχέδιο μου λέτε δεν χρειαζόμαστε. Και κάθε φορά που προβλέπω πω άλλη μια χώρα είναι στα όρια τη διάσωσης μου λέτε όχι, όχι δεν υπάρχει πρόβλημα και φτάσαμε εδώ πέρα στα πρόθυρα τη δεύτερη ελληνικής διάσωση και μου λέτε πως δεν υπάρχει εναλλακτική. Πρέπει να συνεχίσουμε αυτό το δρόμο. Να αγνοήσουμε το ότι τα ισπανικά ομόλογα μα λένε πώ θα ακολουθήσει η Ισπανία. Ε, σε τι χάλι μα φέρατε. Έχετε μέχρι στιγμή 100% λάθος στις προβλέψεις σα για το ευρώ. Και όταν μου λέτε σήμερα πως το πακέτο αυτό θα βάλει την Ελλάδα στον δρόμο της ανάπτυξη, όχι. Θα τη βάλει στον δρόμο της τρίτης διάσωση που θα συζητήσουμε σε λίγους μήνες από σήμερα. Πρέπει να πω πως είναι πραγματικά αειδιαστικό να βλέπουμε τη χώρα που εφήβρε τη δημοκρατία να την κάνετε ό,τι θέλετε εσείς και το αποκρουστικό Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και να μας λένε πως πρέπει να δεχτούν αυτό το πακέτο λιτότητας, να περικόψουν την οικονομία τους σε ένα επίπεδο που θα τους φέρει σε τελείως, σε κατάσταση ύφεσης. Και λένε πως ε, μόνο ο μονεταρισμός είναι λύση. Και βλέπετε οι άνθρωποι τρελαίνονται, βγαίνουν στους δρόμους, υπάρχει βία και μόνο να χειροτερεύσει μπορεί η κατάσταση. Του αφαιρέσατε όχι μόνο τα λεφτά, αλλά και τη δημοκρατία του. Οπότε αυτό το οποίο θα έκαναν οι πραγματικά καλοί Ευρωπαίοι είναι να δώσουν εναλλακτική λύση. Να βοηθήσουν του Έλληνε να έχουν ξανά δικό του νόμισμα. Να του επιτρέψουν την υποτίμηση να αναδιαπραγματευτούν το χρέο του γιατί ο λόγο σε σχέση με το ΑΕΠ έχει περάσει πλέον το σημείο χωρί επιστροφή και τότε μόνο μπορούν να λειτουργήσουν τα πακέτα λιτότητα. Τότε μόνο θα δεχτεί ο ελληνικό λαό αυτέ τι περικοπέ. Εάν συνεχίσουμε την τωρινή πορεία είναι ο δρόμος για οικονομική και κοινωνική καταστροφή. Η κυρία Τζαβέλα, βλέπω ότι ζητάει το λόγο με μπλε δελτίο. Θέλετε να δεχθείτε, παρακαλώ. Κύριε Φάρετς, δέχεστε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Φάραντ αν ξέρει το ύψος του εξωτερικού χρέους της Μεγάλης Βρετανίας και αν πιστεύει ότι μπορεί η Μεγάλη Βρετανία μόνη ως μοναχικό νησί να τα βγάλει πέρα. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Πριν από 20 χρόνια Είμαστε τμήμα του μηχανισμού συναλλάγματος. Ε, προσπαθούσαμε να αντισταθούμε κατά του γερμανικού μάρκου με επιτόκιο διπλάσια από αυτά που θα έπρεπε να είναι. Ε, οι Βρετανοί έχασαν τις θέσει εργασία του και τελικώ βγήκαμε έξω από αυτό το μηχανισμό, ε, έπεσαν τα επιτόκια και ζήσαμε ωραίου καιρού στη διάρκεια τη δεκαετία του 90. Δεν μπορούμε να συγχωνεύουμε διαφορετικέ οικονομίε με διαφορετικά ποσοστά ανάπτυξη, με διαφορετικέ διαδρασμέ παγκοσμίων. Εμεί το μάθαμε το μάθημά μα. Δόξα τω Θεώ δεν ενταχθήκαμε στο ευρώ. Εσείς είστε δυστυχώς παγιδευμένοι σε μια οικονομική φυλακή. Ευχαριστώ. Για 1,5 λεπτό, κύριος Μάντλενερ. Ναι, ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Μπαρόζο μας είπε την ε, Τρίτη πως ε, η Ελλάδα μπορεί να υπολογίζει στην ευρωπαϊκή ε, βοήθεια. Η Ευρώπη θα παρασταθεί, μας είπε. Μα δεν απαγορεύεται σύμφωνα με τη συνθήκη της Λισαβόνας η βοήθεια στην Ελλάδα. Δεν θα πρέπει τα εθνικά κοινοβούλια ένα-ένα να εγκρίνουν αυτή τη βοήθεια και μπορούν να πούν και όχι. Κύριε Πρόεδρε, η δύναμη της Κομισιόν και η εξουσία της συνεχώς εξαπλώνεται. Η Κομισιόν θεωρεί πως μπορεί να κυβερνά όλες τις ευρωπαϊκές χώρες υπό την ηγεσία του κυρίου Μπαρόσο. Και κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Μπαρόσο δεν έχει εκλεγεί δημοκρατικά. Κανένας Ευρωπαίος δεν ψήφισε αυτόν τον άνθρωπο. Μια κυβέρνηση η οποία κυβερνά χωρίς νομοποίηση, ε, μία λέξη περιγράφεται και λέγεται δικτατορία. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε δικτατορία στην Ολλανδία. Είναι απαράδεκτο να αποφασίζει το εάν θα στηρίξει η Ολλανδία την Ελλάδα. Μόνο ένας μπορεί να το κάνει και είναι το Ολλανδικό Κοινοβούλιο. Η δε βοήθεια αυτή είναι άχρηστη, θα βλάψει την Ολλανδική οικονομία γιατί ξέρετε πως ακόμα και αν εξαφανιστεί το ελληνικό χρέος το πρόβλημα δεν θα λυθεί. Οπότε το συμπέρασμα πρέπει να είναι άλλο. Η μόνη μακροπρόθεσμη λύση είναι οι Έλληνες να ξαναφέρουν τη δραχμή, να υποτιμήσουν και να μην ε, αποπληρώσουν ολόκληρο το χρέος. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο πρόεδρος της Επιτροπής έχει το λόγο. Κύριε Βαρόσου. Θα ήθελα να δώσω απάντηση σε δύο συγκεκριμένα ερωτήματα που διατυπώθηκαν απευθυνόμενα προ εμέ. Δεν θέλω να επισταλθώ στην ιδεολογική αυτή συζήτηση για την Ευρώπη, αλλά θα ήθελα να πω ότι είναι ενδιαφέρον το ότι η άκρα αριστερά και η άκρα δεξιά είναι ενωμένε κατά του κατά του ευρωπαϊκού εγχειρήματο. Πολύ ενδιαφέρον θέμα. Για άλλη μια φορά λοιπόν απευθύνω σε όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις της Ευρώπης έκκληση εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και στην Ελλάδα να ενωθούν με συνένεση και να κάνουν ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν για να εξασφαλίσουν ανάπτυξη και ευημερία στην Ευρώπη. Τα δύο συγκεκριμένα ερωτήματα είχαν να κάνουν με τον φόρο των χρηματοπιστωτικών ε, συναλλαγών και τον, ε, τις θέσεις μας για την αντίστροφη ειδική πλειοψηφία. Και θα ήθελα να πω για τον φόρο των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών ότι η πρόταση που θα καταθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά πάσα πιθανότητα τον Οκτώβριο θα έχει να κάνει με φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών κάναμε τη μελέτη αξιολόγησης ε, των επιπτώσεων μπορούσε να υπάρχει ένας φόρος ε, χρηματοπιστωτικών συναλλαγών όπως προτιμούμε έχοντας μελετήσει τις υποθέσεις διότι δεν είναι ισοδύναμος με τον ε, ΦΠΑ. Γι' αυτό λοιπόν την πρότασή μας για το φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών θα την καταθέσουμε τον Οκτώβριο. Για το δεύτερο ερώτημα του κ. Φερχόφστατ. Θέλω να καταστήσω ε, σαφές ότι το, ε, η Επιτροπή είναι υπέρ της αντίστροφης ειδικής πλειοψηφίας. Έχουμε υποστηρίξει τις θέσεις σας ταυτόχρονα και όλη η ΡΕΝ θα έχει την ευκαιρία να σας ομιλήσει σήμερα, αργότερα απόψε. Θα σας απευθύνουμε λοιπόν έκκληση προς το Κοινοβούλιο αλλά και προς το Συμβούλιο για να δούμε αν τελικά μπορούμε να καταλήξουμε σε συμφωνία. Διότι πιστεύουμε επίσης ότι χάρη στις θέσεις του Κοινοβουλίου έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος και στο θέμα του πακέτου διάσωσης, του θέμα του πακέτου που έχουμε τώρα να συζητήσουμε και γι' αυτό ευχαριστώ το Κοινοβούλιο, ιδιαίτερα τους βουλευτές που ασχολήθηκαν περισσότερο με το θέμα αυτό, αλλά και την Ουγγρική Προεδρία που έκανε πολύ σημαντική δουλειά και εν τέλει ευχαριστώ όλους εσάς τους βουλευτές για την υπευθυνότητα που επιδείξατε. Γιατί το κόστος, το τίμημα του να μην συμφωνήσουμε σε αυτό το πακέτο θα είναι πάρα πολύ ψηλό δεδομένων των συνθηκών. Η Επιτροπή είναι υπέρ της κοινωτικής προσέγγισης, είναι υπέρ της όσο πιο φιλόδοξης επιλογής και πιστεύω ότι και εσείς αυτές τις θέσεις πρεσβεύετε. Ευχαριστώ. Ελπίζω να ήταν συγκεκριμένες οι απαντήσεις μου σε μια συγκεκριμένη ερώτηση. Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε. Βέμπερ για δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε του Συμβουλίου, κύριε Πρόεδρε της Κομισιόν, κυρίες και κύριοι, ακούστηκαν ήδη κάποια πράγματα για την Ελλάδα. Δύο σκέψεις θα ήθελα να προσθέσω. Πρώτον, δεν πρέπει να χάνουμε την εξής αρχή από τα μάτια μας τις ε, δύο αρχές δηλαδή οι οποίες ε, αποτελούν χαρακτηριστικά της Ευρώπης. Αφενός η αλληλεγγύη, αφετέρου η ατομική ευθύνη. Θα πρέπει λοιπόν να επιδείξουμε αλληλεγγύη και να δράσουν με ευθύνη οι Έλληνες και από την άλλη μιλήσαμε για τη μεγάλη δοκιμασία την οποία περνάει η Ευρώπη και για το ότι θα μπορούσε να αποτύχει και να ξαναξυπνήσουν παλαιά ε, δαιμόνια στην Ευρώπη. Δεν πρέπει να μιλάμε μόνο για τα προβλήματα αλλά και για τις επιτυχίες, ε, για το ότι πώς κατάφεραν να βγουν από την κρίση οι χώρες Βαλτικής, πώς η Ιρλανδία του χρόνου με την ευρωπαϊκή στήριξη θα καταφέρει να επιστρέψει στις ε, αγορές. Οπότε έχουμε μια απόδειξη για το ότι ενωμένοι είμαστε ισχυρότεροι από ό,τι μόνοι μας. Κυρίες και κύριοι. θα πρέπει να αναφερθούμε και στο άλλο βεβαίως ε, κορυφαίο θέμα της ε, Συνόδου, την ε, μετανάστευση, αλλά και στη Σέγγεν έχουμε την ίδια κατάσταση, δηλαδή μια μεγάλη κατάκτηση της Ευρώπης καταστρέφεται από τους εθνικούς εγωισμούς. Είδατε πως έφτασαν 18.000 πρόσφυγες στην Ιταλία αλλά ξέρουμε πως αυτό δεν είναι ιδιαίτερη επιβάρυνση για την Ιταλία. Οι διπλάσιοι βρίσκονται στο Βέλγιο, οπότε δεν είναι σωστή η Ιταλική αντίδραση και ήταν αυτό εσωτερική πολιτική και αφορούσε τον Υπουργό Εσωτερικών, τον ε, κύριο Μπόση αυτό το οποίο έγινε. Και στην Δανία και αλλού πάλι οι λόγοι για αυτές τις δράσεις ήταν η εσωτερική πολιτική. Γι' αυτό ζητώ από το Συμβούλιο να στείλει ένα σαφές μήνυμα. Όταν μιλάμε για τη μετανάστευση και για τη Σέγγεν θα πρέπει οι κυβερνήσεις να στείλουν ένα διαφορετικό μήνυμα και να πούν πως δεν θέλουμε εθνικούς εγωισμούς και σε αυτό το θέμα αλλά θέλουμε να υπερασπίσουμε τη μεγάλη επιτυχία της ελεύθερης διακίνησης στην Ευρώπη. Και κύριε Πρόεδρε της Κομισιόν έχετε οπωσδήποτε τη στήριξη του Κοινοβουλίου γι' αυτό. Ευχαριστώ κύριε Βέμπερ. Ο κύριος Σόμποντα. Δύο λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε του κύριε Πρόεδρε Τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ήθελα καταρχά να φερθώ σε ένα θέμα που με ενδιαφέρει ιδιαίτερω και είναι η Κροατία φυσικά. Ελπίζω το ταχύτερο δυνατό να καταλήξουν οι συζητήσει με την Κροατία έτσι ώστε να ενταχθεί όσο δυνατόν πιο νωρί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Ο κύριο Φιούλε αλλά και ο ίδιο ο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ουγγρική Προεδρία εν προκειμένου έχουν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και νομίζω ότι αποτελεί αυτό ένα πάρα πολύ καλό και σημαντικό μήνυμα και δείγμα για το πώ μπορούν χώρε οι οποίε ταλανίζονται από προβλήματα προβλήματα και κρίσεις όπως τα Βαλκάνια ε, να αντιμετωπίσουν σωστά τα προβλήματά τους. Αντιμετωπίζουν λέω και όχι επιλύουν γιατί δεν έχουν επιλυθεί όλα τα προβλήματα. Υπάρχουν κάποια ζητήματα στα οποία βλέπουμε πολύ σοβαρά προβλήματα ακόμη και απαράδεκτη κατάσταση, αλλά κατά βάση να έχουν αντιμετωπίσει τα σοβαρότερα ζητήματα. Επιτρέψτε μου τώρα να δύο λόγια για την Ελλάδα. Κύριε Πρόεδρε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι δύσκολο να εξηγήσουμε στου πολίτε το γιατί δεν μπορούμε να δώσουμε μια λύση φερρυπίν για το πακέτο τη οικονομική διακυβέρνηση. Αλλά θα είναι δύσκολο, κύριε Πρόεδρε τη Επιτροπή, να εξηγήσουμε στου πολίτε και γιατί μπορεί να επικεντρωνόμαστε μόνο σε μέτρα λιτότητα. Εδώ γίνεται λόγο για την ανάπτυξη. Εννοούμε ότι χρειάζεται κάτι που θα βοηθήσει την ανάπτυξη. Τι μπορεί να είναι αυτό. Δεν μπορεί να είναι βέβαια το να πιστεύουμε ότι η λιτότητα ε, οδηγεί σε ανάπτυξη και μόνο η λιτότητα. Δεν μπορεί αυτό να είναι μια απάντηση και σα διαβεβαιώ ότι αυτό δεν είναι αριστερή επιλογή. Και στην εφημερίδα Λεμόντα ακόμη χτε, που δεν είναι καθόλου αριστερό φίλο, ε, γινόταν ε, σχόλια του τύπου Ναι, χρειάζεται η λιτότητα, αλλά δεν αρκεί, χρειάζεται και ε, ανάπτυξη. Για την ανάπτυξη δεν χρειάζονται επενδύσει. Και βέβαια είναι το θέμα των ιδιωτικοποιήσεων ε, εντωμεταξύ. Ξέρετε ότι η Ελλάδα θα πρέπει να προχωρήσει ταχύτατα σε ιδιωτικοποίηση, αλλά αν αυτό γίνει με υπερβολικά στενά χρονικά όρια, θα, είναι, θα καταρρεύσει το σύστημα, θα είναι ε, άχρηστες αυτές οι ιδιωτικοποίησεις δεν θα φέρουν έσοδα όπως είπε και ο κύριος Μπίση και θα γίνουν δωρεάν. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να τις κάνουμε τις ιδιωτικοποίησεις κατά τρόπο οργανωμένο και τέτοιο ώστε να φέρουν πραγματικά έσοδα και να γίνουν με σωστούς όρους. Φερρυπίν με ένα ταμείο υποστήριξης ε, της ιδιωτικοποίησης Φερρυπίν με κάποια μέσα οικονομικά που θα μπορούσαν να στηρίξουν την Ελλάδα σε αυτή τη πορεία. Κύριε, Επίτροπη, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, εμείς είμαστε υπέρ της ε, αυστηρής δημοσιονομικής πολιτικής, υπέρ της δημοσιονομικής πειθαρχίας, όχι ε, υπέρ των υπερβολικών δαπανών. Αλλά η υπερβολική και άκρα λιτότητα ούτε, ούτε την Ελλάδα πρόκειται να, να σώσει, ούτε τις τράπεζες πρόκειται να διασώσει, ούτε το φορολογούμενο πρόκειται να βοηθήσει θα καταρρεύσουν τα πάντα και γι' αυτό χρειάζεται και πέραν των ρυθμιστικών μέσων ανάπτυξη. Ανάπτυξη, απασχόληση που έχουν καθοριστική σημασία για το μέλλον τη Ελλάδα και ολόκληρη Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριο Ράνστορ ζητάει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, έχω μία ερώτηση προς τον κύριο Σπόμποντα. Συμφωνείτε με την άποψη ότι σε κάποια κράτη-μέλη χρησιμοποιείται η κρίση ως μέσο για μια αργή και λανθάνουσα ιδιωτικοποίηση, εξαγορά ουσιαστικά της ιδιοκτησίας ε, σε όλα τα κράτη που αντιμετωπίζουν κρίση υπάρχουν ουσιαστικά προβλήματα. Δεν υπάρχει λόγος ε, να συγκαλύπτουμε την κατάσταση. Χρειάζεται να δοθούν λύσεις και όταν κάποιες ε, ε κάποιοι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας ε, σπρώχνουν τις χώρες ε, αυτές στο χείλος του γκρεμού μπορεί να καταρρεύσουν. Αυτό είναι βέβαιο. Από την άλλη βεβαίως δεν ε, είναι σωστό ότι θα πρέπει να ε, αρνηθούμε κάθε εξέλιξη, ιδιωτικοποίηση κτλ. Και πιστεύω ότι η κυβέρνηση Παπανδρέου κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Θα πρέπει να τη στηρίξουν τα συνδικάτα και να την αφήσουν να προχωρήσει προ μια σωστή πολιτική, μια πολιτική που θα αναπτύξει, που θα επιτρέψει την ανάπτυξη τη χώρα. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει θέμα κατάχρηση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ευχαριστώ. Κύριο Λάμπστορφ έχει το λόγο. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε μετά την ψήφο εμπιστοσύνη χθε στην Αθήνα με το αποτέλεσμα που ξέρουμε η εφημερίδα Bild στη Γερμανία είχε τίτλο ο Παπανδρέου επέζησε η Ευρώπη ανασένει και εγώ χάρηκα αλλά τώρα για να ανασάνω είναι πάρα πολύ νωρίς το θέμα είναι την επόμενη εβδομάδα να περάσει το μεγάλο πακέτο λιτότητας. Και ακόμα τότε δεν μπορούμε να ανασάνουμε. Θα πρέπει να ακολουθήσουν και άλλα πολλά βήματα και μέτρα μέχρι να ξεπεραστεί η κρίση. Πιστεύω πως αυτό το οποίο υπόθηκε είναι σωστό. Οι άνθρωποι στην Ελλάδα πράγματι χρειάζονται και ένα μήνυμα θετικό, αλλά και φω στο τέλο του τούνελ θέλουν και οι άνθρωποι που δίνουν τα χρήματα. Γιατί έχουν την αίσθηση πω δίνουν, δίνουν, δίνουν και δεν γίνεται τίποτα. Στην Ελλάδα δεν έχουν την αίσθηση ότι κόβουμε, κόβουμε, κόβουμε και πάλι δεν γίνεται τίποτα. Οπότε ναι εντάξει η ιδιωτικοποίηση, ναι να απελευθερωθεί αυτή η απολυθωμένη οικονομία, αλλά θα πρέπει να προχωρήσει και η χώρα αυτή προς τα μπρος και να στηρίξει και η Νέα Δημοκρατία. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει από τον κύριο Σαμαρά. Πράγματι θα πρέπει να βοηθήσουμε και με τα κονδύλια τα οποία δεν χρησιμοποιούνται τα ευρωπαϊκά, όπω είπε και ο κύριο πρόεδρο τη Κομισιόν, και από την ανάπτυξη δεν αποφελήθηκαν μόνο οι Έλληνε, αλλά ολόκληρη η Ευρώπη. Πρέπει να ενισχυθεί επίση το σύμφωνο σταθερότητα, να εμποδίσουμε μελλοντικέ κρίσει και σε αυτό βεβαίω. Οπωσδήποτε ανήκει αυτή η αντίστροφη δική πλειοψηφία, η οποία βεβαίω σε ένα απλόν άνθρωπο δεν λέει απολύτω τίποτα. Γιατί αν γίνει αυτό πραγματικά θα δείξουμε εάν έχει δόντια και ουσία το σύμφωνο σταθερότητας ή όχι. Γι' αυτό υποστηρίζουμε ακριβώς την αντίστροφη αυτή ειδική πλειοψηφία στην προληπτική φάση του συμφώνου. Είναι ξεκάθαρο για εμάς ε, κύριε Μπαρόσο και χαιρόμαστε που έχει την ίδια άποψη η Κομισιόν και θα σας στηρίξουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Λάμσδορφ. Η κυρία Τζαβέλα για ένα λεπτό. Κύριε Λάμπστορφ, θα δεχτείτε μια ερώτηση από τον κύριο Γκίγκολτ. Εγώ, κύριε Λάμπστορφ, συμφωνώ μαζί σας πως χρειάζεται πολιτική ενότητα επιγόντως στην Ελλάδα, αλλά αυτό θα πρέπει να ξεκινήσει με το να γίνουν επιτέλους δίκαιες προτάσεις. Ενότητα στη χώρα θα υπάρχει μόνο όταν υπάρχει εμπιστοσύνη στις πολιτικές και οικονομικές ελίτ και αυτό σημαίνει πως οι προτάσεις αυτές θα πρέπει να οδηγήσουν στην ενότητα. Αλλά εγώ θέλω να θέσω το εξή ερώτημα. Θα ήθελα να υπάρχει ενότητα και στην ομάδα σας. Ζητάτε ευρωομόλογα. Στη Γερμανία λέτε τα ευρωομόλογα είναι κατάρα. Στην ομάδα σας, στην Ομοσπονδιακή Γερμανική Βουλή, είχατε λάβει θέση κατά κάτι, κάποιες τέτοιες Μα ο Πρόεδρος, Κύριε Γκίγκολτ, πρέπει να κάνετε ερώτηση, όχι δηλώσεις με την μπλε κάρτα. Οπότε δεν έχει να απαντήσει τίποτα ο κύριος Λάμσδορφ. Η κυρία Τζαβέλα για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, ω Ελληνίδα θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για όλη τη στήριξη που έχει παράσχει στην Ελλάδα μέχρι τώρα ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εργαζόμενους στην επιτροπή που 18 μήνες τώρα δουλεύουν πολύ σκληρά για την επίλυση της ελληνικής κρίσης. Κυρίες και κύριοι, μιλήσαμε πολύ σε αυτό το Ευρωκοινοβούλιο σήμερα για την Ευρώπη. Θα ήθελα μόνο ένα σχόλιο να κάνω πατριωτικού περιεχομένου σε αυτό το πολυεθνικό ακροατήριο. Την Ευρώπη εμείς οι Έλληνες την ονομάσαμε Ευρώπη και συμβάλαμε αποφασιστικά σε αυτό που λέμε ευρωπαϊκός πολιτισμός και ευρωπαϊκές αρχές. Τι ζητάμε οι Έλληνες πολιτικοί και ο ελληνικός λαός. Ζητάμε το σεβασμό σας και την αλληλεγγύη σας. Τι μπορούμε να υποσχεθούμε. Ότι θα δουλέψουμε πολύ σκληρά για να ορθοποδήσει η χώρα την οποία εμείς οι ίδιοι και πρώτα απ' όλα εμείς έχουμε το πρόβλημα και την ενοχή τη φτάσαμε εκεί. κύριε πρόεδρε τρεις προτάσεις επιτρέψτε μου. το πρώτο βήμα ένα λεπτό κύριε πρόεδρε μπορώ. τρεις προτάσεις πολύ γρήγορα. ευρωπαϊκό Κυρία Τζαβέλα, είχατε ένα λεπτό χρόνο ομιλία. Το έχετε ξεπεράσει εδώ και πολλή ώρα. Λοιπόν, Το λόγο έχει ο κύριο Μπρόν τώρα για ένα μισή λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, η Προεδρία πολλών ετούντων άσυλο από τη Λιβύη και από την Τινουσία θα βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη. Η Τινουσία είναι μια χώρα που εκδίωξε τον ε, δικτάτορα από πού φεύγουν λοιπόν αυτή την ίση ε, από τη δημοκρατία. Ο κύριος Μπεναλή ε, ε, μπορεί να είναι και στο τέλος της ουράς. Ε, δεν έχουν γίνει αιτούντε άσυλο αυτοί οι άνθρωποι γιατί ζουν σε μια επικίνδυνη χώρα. Κάτι πρέπει να υπάρχει που να θέτει σε κίνδυνο τη ζωή αυτού του συγκεκριμένου ανθρώπου. Το θέμα είναι κατά πόσον η Ιταλία και η Μάλτα θα πρέπει να δεχτούν την ε, αίτησή τους γιατί είναι η πρώτα χώρα στην οποία θα καταφτάσουν ε, και αν θα πρέπει να δεχτούν και τη συμφωνία οι υπόλοιπε χώρε. Ε, η άποψή μου είναι ότι δεν θα πρέπει να το δεχτούμε και αργά ή γρήγορα πρέπει να επιστρέψουν στη Βόρεια Αφρική. Το να ζητά κάποιο άσυλο και να θεωρείται απαραίτητο προπόθεση για να το δεχτούμε θα πρέπει να πάψει να ισχύει. Θα πρέπει τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση αν πρέπει να αρνηθεί διεθνείς συμφωνίες να το κάνει. Έφτασε η στιγμή να σταματήσει η ροή των μετανιστών και να τους δείξουμε το δρόμο προς την επιστροφή. Η ένταξη της Κροατίας επίσης θα συζητηθεί. Τι μέτρα θα λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να διασφαλίσει ότι θα γίνει ένα δίκαιο δημοψήφισμο που θα ε, επιτρέψει να εισακουστούν και οι δύο πλευρές και ε, δεν θα υπάρξει και κατασπατάληση χρημάτων. Φαντάζομαι ότι ένα ελεύθερο και δίκαιο δημοψήφισμα δεν βρίσκεται στα χαρτιά. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι είναι κατά της Κροατίας και δυστυχώς δεν θα τους επιτραπεί να υψώσουν τη φωνή τους. Ευχαριστώ κύριε Μπρόντς. Και τώρα η κυρία Γκάλ Πέλτς για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η προσοχή συνεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα πρέπει να εμπνέει δικαιοσύνη, και εμπιστοσύνη. Πρόκειται για μια στιγμή ιστορική. Ιστορική γιατί θα πρέπει να εντοπιστούν, να αποκαλυφθούν οι μεγάλε προκλήσει που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και να δοθούν οι σωστέ απαντήσει. Οι απαντήσει όμω όλε είναι ανελέγχοντε μεταξύ του. Και επιτρέψτε μου καταρχά να ευχαριστήσω θερμά την Ουγγρική Προεδρία για την πολύ καλή δουλειά που έχει κάνει και ιδιαιτέρω την κυρία Γκέρι υφυπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, η οποία ε, ήταν σε αυτό το εξάμεινο πανταχού παρούσα. Έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά. Η Ουγγρική Προεδρία έχει τηρήσει το πρόγραμμά της και έχει ακολουθήσει μια στάση θετική, πολύ θετική και ανοιχτή προς το Κοινοβούλιο. Έτσι λοιπόν ε, υπάρχουν μεγάλα, ε, μεγάλες προκλήσεις για ολόκληρη την Ευρώπη Έχουμε την νέα οικονομική διακυβέρνηση με τα έξι προτάσεις που αποτελούν μεγάλη πρόκληση. Ένα σύνολο νομοθετικό στο οποίο παραμένουν ακόμη εκρεμή κάποια ζητήματα και στο οποίο έχουν, φέρουν τεράστια μέρος ευθύνη στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Φέρουν ευθύνη να ε, ε, λάβουν αποφάσεις, να συμφωνήσουν δηλαδή για να προχωρήσουμε στο μέλλον με σαφείς κανόνες για την ε, μοίρα του Συμφώνου και Σταθερότητας, τη διατήρησή του δηλαδή ή αλλιώς την αντιμετώπιση των ζητημάτων μέσα από διμερείς συμφωνίες και μια νέα προσέγγιση στο θέμα της οικονομικής κυβέρνησης με κοινούς ευρωπαϊκούς κανόνες, κοινέ ευρωπαϊκές προσεγγίσεις που θα ενισχύσουν τον, που θα επιτρέψουν ταυτόχρονα και την ενίσχυση του συντονισμού, του οικονομικού συντονισμού και την ανάπτυξη μιας ισχυρής Ευρώπης. Αυτό αναμένει ο πολίτη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Περιμένει κοινού κανόνε. Κοινού κανόνε που θα εφαρμόζονται κατά τρόπον ο οποίο θα εξασφαλίσει και την σταθερότητα του κοινού νομίσματο αλλά και την προστασία του πολίτη από τι συνέπειε τη κρίση. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Ο κύριος Λόπες Αγγιλάρ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι η συζήτηση είναι για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα γίνει στις 23 και 24 Ιουνίου και εξακολουθεί να επικεντρώνεται στην ε, σημαντική οικονομική κρίση, στα προβλήματα του ευρώ και στην Ελλάδα αλλά να σας πω ότι ε, δεν εξαντλείται εκεί η ημερήσια διάταξη. Πρέπει να συζητήσουμε και ε, στοιχεία τα οποία αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων και πιο συγκεκριμένα τη Σέγγεν, που είναι ο βασικός ε, μοχλός που επιτρέπει την ελεύθερη μετακίνηση ανθρώπων. Και δεν θα πρέπει μετά από τη δημοκρατία στη Βόρεια Αφρική να μην δώσουμε μία σαφή απάντηση στα θέματα αυτά. Μπορεί να πρέπει να μεταρρυθμίσουμε τη Σέγγεν όπως λένε κάποιοι. Όχι, το αντίθετο. Θα πρέπει να την ενισχύσουμε τη Σέγγεν. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι μας λένε ότι ε, αν έχουμε αναπέντεχες μεταναστευτικές ροές όπως έγινε στα Κανάρια νησιά στην Ισπανία το 2004 και το 2006 η απάντηση δεν θα πρέπει να είναι απλώς ε, περισσότερη και καλύτερη Ευρώπη αλλά και μια συνεισφορά με αλληλεγγύη στο αίτημα για περισσότερη δημοκρατία για τις γείτονες χώρες. Γνωρίζουμε ότι η Μάλτα, η Ιταλία και η Γαλλία έζησαν αντίστοιχε πιέσει. Αλλά θα πρέπει και το Συμβούλιο να συνεισφέρει να συμπληρώσει το πακέτο του ασύλου, να συμπληρώσει το πακέτο της μετανάστευσης, να συμπληρώσει τη μεταρρύθμιση του κανονισμού Frontex και να θέσει σε εφαρμογή τη ρήτρα λιδεγγύης που αναφέρεται στο άρθρο 80 της Συνθήκης Λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης που σημαίνει εφαρμογή της Οδηγίας 2001-55. Επίσης θα ήθελα να εκφράσω και την ανησυχία μου για το μήνυμα το οποίο διαβιβάστηκε για την δημιουργία ενός μηχανισμού απάντησης που επιτρέπει να ε, χρησιμοποιήσουμε εκ νέου τα εσωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκή Ένωση σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης. Θα πρέπει να γνωρίζουμε γιατί ακριβώς μιλάμε και ποια θα πρέπει να είναι η σαφής ενωσιακή ε, ευρωπαϊκή διάσταση για να μην είναι αντιπαραγωγική. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η κυρία Βάλεν για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Μετά από ένα έτος ενθουσιασμού και ανοχής για την Ευρώπη βλέπουμε μετά από πολλά τέτοια χρόνια μια επιδείνωση του κλίματος ακόμα και εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ζητήματα όπως η ελεύθερη διακίνηση, η μετανάστευση και πάνω απ' όλα βεβαίως τα λεφτά. Δυστυχώς η παγκόσμια αυτή οικονομική κρίση τονίζει τις χειρότερες εθνικιστικές και λαϊκιστικές απόψεις. Ε, το χάος που δημιουργείται κάθε μέρα από τις δηλώσεις ε, για την Ελλάδα εντείνει την σύγχυση και δημιουργεί περισσότερη κερδοσκοπία στις αγορές ε, και κίνδυνο πραγματικό για μετάδοση και στα άλλα κράτη-μέλη. Η Ευρώπη σηκώνει το βάρος της ευθύνης της και το ίδιο κάνουν και οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Εάν ε, είχε γίνει αυτό πριν από ένα έτος δεν θα περνούσαμε από το ένα σχέδιο διάσωσης στο άλλο. Τώρα χρειαζόμαστε όχι άλλες τεχνικές λύσεις αλλά συνοχή, αποφασιστικότητα και ενότητα γιατί ε, βρισκόμαστε σε έναν ψυχολογικό πόλεμο και αυτό το οποίο δοκιμάζουν βεβαίω οι αγορές είναι η ευρωπαϊκή ενότητα και όχι η ελληνική λιτότητα. Θα πρέπει λοιπόν να στείλουμε ένα μήνυμα ενθαρρυντικό ότι η Ευρώπη στηρίζει την Ελλάδα και πλέον πρέπει να μειώσουμε το επιτόκιο και να δείξουμε μεγαλύτερη ευελιξία στην πρόσβαση στα ευρωπαϊκά κονδύλια. Επιπλέον η Ελλάδα θα πρέπει και αυτή να πάρει τις μοίρες της, τη μοίρα της στα χέρια της. Οι μεταρρυθμίσεις είναι απαραίτητες, αλλά βεβαίω η λιτότητα από μόνη της δεν οδηγεί στην ανάκαμψη. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε στα βασικά επενδύσεις και ανάπτυξη. Ελπίζω αύριο κανείς Ευρωπαίος ηγέτης να μην σταματήσει τις πληρωμές της αλληλεγγύης. Γιατί βεβαίως πρόκειται για την Ευρώπη που κρίνεται. Αν παραστεκόμαστε στην Ελλάδα, παραστεκόμαστε στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ, Μποργέτσιο, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για την Ελλάδα νομίζω ότι αρκεί να ακούσαμε τα όσα συζητήθηκαν εδώ για να καταλάβουμε σε τι σημείο βρίσκεται η ευρωπαϊκή διακυβέρνηση. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα ανασαφή κατάλογο χωρίς συγκεκριμένους στόχους. Δεν ακούσαμε τίποτα ε, για κάτι συγκεκριμένο και αν εγώ ήμουν ένας Έλληνας εργαζόμενος ή ένας μικροεπιχειρηματίας ο οποίος ε, οδεύω προς τη πτώχευση να είχα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι μου μετανάστευση. Άκουσα να επικρίνεται η Ιταλία γιατί δεν θέλει να υποδεχτεί τους μετανάστες. Αλλά η κυρία Μάλστρομ πριν από λίγες ώρες έκανε μια δημόσια δήλωση και είπε ότι όταν ξεκίνησε η τραγωδία από τη Λιβύη ε, όλοι δεσμεύθηκαν να υποδεχθούν τουλάχιστον 500 πρόσφυγες ανά χώρα στην πράξη δεν τους υποδέχθηκε κανείς. Ε, υπάρχει και η περίπτωση της Νορβηγία, ε, Εκφορτώνονται στη Λαμπεντούζα ε, και τους αναλαμβάνουμε μόνο εμείς. Η Ιταλία τους υποδέχθηκε. Η Ιταλία επαναλαμβάνω. Αναφερθήκατε στον Υπουργό Μπόση, υπάρχει και ο υπουργό Εσωτερικών, ο οποίος δεν ανήκει στη Λίγα του Βορρά και που και πάλι τους υποδέχθηκε. Τέλος, το κεφάλαιο Κροατία πολύ σημαντική η προσχώρηση της Κροατίας, αλλά θα πρέπει να υπενθυμίσουμε και αυτό που είπε ο Πάπας στους Κροάτες. Προσέξτε, πρόκειται για ένα γραφειοκρατικό και κεντροκρατικό σύστημα. Ευχαριστούμε κύριε Μποργέτσιο. Για δύο λεπτά ο κύριος Μάουρο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η πολυπλικότητα της ημερήσιας διάταξης ε, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Μα φέρνει αντιμέτωπου με την έλλειψη μέσων που έχουμε στη διάθεσή μα. Τι έχουμε, έχουμε στη διάθεσή μα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή ένα οικοδόμημα εν εξελίξη που δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί και που πολλές φορές το γεγονός ότι είμαστε τόσο ευάλωτοι και τόσο φοβισμένοι δεν μας επέτρεψε να το ολοκληρώσουμε. Έχουμε στη διάθεσή μας την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν έχουμε στη διάθεσή μας τις ΗΠΑ της Ευρώπης. Δεν έχουμε δηλαδή ένα μέσο το οποίο ε, όταν υπάρχει ε, μια κυβέρνηση που αμφιταλαντεύεται και που ε, συνδέονται οι αποφαταλαντεύσεις αυτές με εσωτερική λογική, δεν μπορεί να οδηγήσει στη λύση των προβλημάτων. Για να μπορέσουμε να έχουμε λοιπόν στη διάθεσή μας τις Ηνωμένε Πολιτείε της Ευρώπης, πρέπει να υπάρχει μια ηγεσία που να είναι ε, αυτή η οποία θα προέρχεται από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ιδίω από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Νομίζω, λείπει ο κύριος Μπαρόζο, ότι το γεγονό ότι ήταν τόσο επιφυλακτικό ε, του έδωσε εισάξια την ε, δεύτερη του θητεία. Εάν λοιπόν τη δεύτερη φορά εξελέγει για την ε, ε, ταπεινοφροσύνη του, την επόμενη φορά θα ήθελα να τον εκλέξουμε για το σθένος του, για το θάρρος που πρέπει να επιδείξει. Σε αυτή λοιπόν την ημερήσια διάταξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να πείσουν τις εθνικές κυβερνήσεις να προτάξουν τα δικά, τους, τα δικά μας πριν από τα κοινά τους συμφέροντα. Αλλιώς θα συνεχίσουμε να κάνουμε συζητήσεις όπου θα ε, λέμε ότι δυστυχώς για εσωτερικούς λόγους η γαλλική κυβέρνηση ανέλαβε πρωτοβουλία για τη Σέγγεν, η ιταλική κυβέρνηση αρνήθηκε να υποδεχθεί το δεν ξέρω ποιον, η ελληνική κυβέρνηση είναι ακόμα πολύ εύθραυστη και δεν μπορεί να αναλάβει τις ευθύνες ε, των επιλογών της. Αλλά το πρόβλημα μας έγκυται αλλού. Χωρίς να διευκρινίσουμε την πολιτική φύση του ευρωπαϊκού προγράμματος, δεν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματά μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Μάουρο. Η κυρία Ποδηματά έχει το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου πρώτα απ' όλα να προσθέσω κι εγώ στις ευχαριστίες που εξέφρασε η συνάδελφος η κυρία Τζαβέλα και θέλω να την ευχαριστήσω γι' αυτό τις ευχαριστίες και προς τα κοινοβούλια και τους λαούς της ευρώπης για την υποστήριξη που έδωσαν και συνεχίζουν να δίνουν στη χώρα μου. η ελλάδα κύριε πρόεδρε κυρίες και κύριοι όπως απέδειξαν και οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών είναι αποφασισμένη να συνεχίσει και να επιταχύνει τις προσπάθειες για δημοσιονομική εξυγίανση και για προώθηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. υπάρχουν όμως για να στεφθούν οι προσπάθειες αυτές με επιτυχία δύο προϋποθέσεις η πρώτη προϋπόθεση είναι να είμαστε σε θέση να δώσουμε στους πολίτες εκτός από τη λιτότητα και μια προοπτική θετική μια προοπτική ανάπτυξης μια προοπτική απασχόλησης μια προοπτική δημιουργίας θέσεων εργασίας. η δεύτερη προϋπόθεση είναι ένα περιβάλλον ασφάλειας και υποστήριξης από την πλευρά της ευρωπαϊκής ένωσης ένα περιβάλλον πολιτικής συνοχής γιατί σε όλη τη διάρκεια της κρίσης αλλά ιδιαίτερα τις τελευταίες εβδομάδες παρακολουθήσαμε και παρακολουθούμε έναν άτυπο δημόσιο διάλογο μεταξύ ευρωπαϊκών πρωτευουσών της ευρωπαϊκής επιτροπής της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας με μια ιδιότυπη επιδιαιτησία από την πλευρά των οίκων αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας σε ό,τι αφορά την περίφημη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στο νέο πακέτο διάσωσης της ελληνικής οικονομίας. και θέλω να πω αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητές συνάδελφοι ότι αυτή η ιδιότυπη επιδιαιτησία δεν τιμά ούτε την ευρωπαϊκή ένωση ούτε την πολιτική. πρέπει να τεθεί ένα τέλος σε αυτήν την κακοφωνία γιατί μόνο μέσα σε ένα περιβάλλον πολιτικής συνοχής θα μπορούμε να ελπίζουμε ότι οι πολύ σκληρές προσπάθειες που καταβάλει ο ελληνικός λαός έχουν τις προϋποθέσεις να στεφθούν με επιτυχία. ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Ποδηματά και κυρία Λάτφορτ τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το κύριο ερώτημα που θα αντιμετωπίσουν αύριο οι Ευρωπαίοι ηγέτε είναι εάν μπορούν να αρθούν στο ύψο των περιστάσεων και να σώσουν την ζώνη του ευρώ και την ελεύθερη διακίνηση στην Ευρώπη χρειάζεται σε περιπτώσεις όπως αυτή να μπορεί κανείς να λαμβάνει τις σκληρές αποφάσεις και χαίρομαι για τις ε, απερίφραστες δηλώσεις του κυρίου Μπαρόσο σήμερα που δεν τις ακούσαμε βέβαια το Μάιο γιατί το Μάιο θα έπρεπε να είχε τραβήξει αυτή της Ιταλίας και της Γαλλίας όπως έκανε τώρα νωρίτερα ο κύριος Βέμπερ ο συνάδελφος. Ο κύριος Μόντι έκανε μια δήλωση στις Financial Times όπου δήλωνε την ε, λύπη του για την ε, μεγάλη ε, υποχωρητικότητα εναντί των μεγάλων κρατών μελών και την υπερβολική ευγένεια που χαρακτηρίζει συνεδριάσεις όπου ο καθένα από τα κράτη-μέλη, το καθένα από τα κράτη-μέλη αποφεύγει να επικρίνει το άλλο σε τέτοιε περιπτώσει. Αυτό σημαίνει κράταμε να σε κρατών να ανεβούμε στο βουνό ουσιαστικά. Η κόρα κασκορά κομμάτι δεν βγάζει. Θα πρέπει να είμαστε σε θέση να καταγγέλουμε τα προβλήματα και γιατί χωρί να είμαστε απόλυτα ειλικρινεί ο με τον άλλον δεν μπορούμε να έχουμε και απόλυτη εμπιστοσύνη. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ο κύριος Προβέρα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μετανάστευση. Είδαμε ότι καμία χώρα δεν μπορεί μόνη της να αντιπατοποιήσει τις μεταναστευτικές ροές. Πρέπει να υπάρχει λοιπόν μια πολιτική διαχείριση των μεγάλων μεταναστευτικών ροών η οποία θα ε, συνδυαστεί με τις πολιτικές ανάπτυξης και θα περιλαμβάνει διμερείς και πολυμερείς συμφωνίες με τις χώρες καταγωγής των μεταναστών. Δυστυχώ, όπως διαπιστώνει η Ιταλία αυτή τη στιγμή, τα μέσα που έχουμε για εξωτερική δράση δεν χρησιμοποιήθηκαν βάσει του πνεύματος ε, των συνθήκων. Τα κράτη-μέλη στην πρώτη γραμμή αναγκάστηκαν ε, να αντιμετωπίσουν την κατεπίγουσα κατάσταση των ε, ε, μεταναστών και των προσφύγων χωρίς να μπορούν να βασιστούν στην Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη. Θα ήθελα να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει σε ποιες περιπτώσεις θα μπορούμε να μιλάμε για μαζική ροή μεταναστών εντός εισαγωγικών βάσει του άρθρου για την προσωρινή μετανάστευση καθορίζοντας σαφή και μετρήσιμα κριτήρια τα οποία να μπορούμε να θεωρήσουμε ως σταθερά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να υπάρχει μια αποτελεσματική κοινή πολιτική για τα θέματα της μετανάστευσης και να υπάρχει ισοκατανομή των βαρών. Ευχαριστώ για δύο λεπτά ο κύριος Σοντή. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ Προεδρεύουσα του Συμβουλίου, θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου προς το πρόσωπό σας και προς την Προεδρία σας και να χαιρετήσω τη στάση της ΕΕ στην Για την Ελλάδα, Καταρχάς, θα θέλω να πω ότι θα πρέπει να εξηγιανθεί η οικονομία και να δοθούν ε, λύσεις προς την ανάπτυξη. Η εξηγένση της οικονομία δείχνει ότι είναι πολύ δύσκολο να διακυβερνά κανείς ε, με το βάρος του παρελθόντος, στραμμένος όμως προς το ε, μέλλον. Θα έλεγα λοιπόν ότι θα έπρεπε να συσταθεί ένας θεσμός διαμεσολαβητή του δανείου ε, ή μάλλον του χρέους έτσι ώστε να είναι σε θέση να προσφέρει αυτός κάποιες λύσεις και ιδέες για τη διαχείριση του υπερβολικού ελλείμματος και του χρέους ε, για να, ώστε να μην υπάρχουν απώλειες από κεφάλαια και να περιοριστεί το χρέος της Ελλάδας έτσι ώστε να μπορούν οι κυβερνήσει να κοιτάξουν προς το μέλλον. Την αναδιάρθρωση που είναι στραμμένη προς το παρελθόν την αναλαμβάνει ο διαμεσολαβητής. Φυσικά θα χρειαστεί και συμμετοχή των τραπεζών που έχουν ε, τεράστια κέρδη. Όταν αγόραζαν το, ε, την προοπτική του χρέους με 16% επιτόκιο, ενώ όταν αυτό έφτασε στο 8% είχαν ουσιαστικά διπλάσιο κέρδος και νομίζω θα πρέπει να γίνει μια διερεύνηση της κατάστασης και του ρόλου που έχουν διαδραματίσει οι οικονομικοί αυτοί φορείς και ιδιαίτερα οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, οι οποίοι οργανισμοί κατά κάποιο τρόπο έκαναν καταχρηστική υποστήριξη και ενίσχυση του χρέους, όπως λέμε στο γαλλικό δίκαιο, δηλαδή ενίσχυσαν τις συνθήκες αυτής της κρίσης και αποκόμισαν και όφελος από αυτήν. Για δε την ανάπτυξη θέλω να υποστηρίξω τις προτάσεις προτάσεις του κυρίου Μπαρόσου, του κυρίου Προέδρου για την χορήγηση ενός δισεκατομμυρίου ευρώ και ένα πραγματικό σχέδιο για ανάπτυξη της Ελλάδας και δεν θα θέλει να υποστηρίξω τις προτάσεις του κυρίου Κονμπεντίτ που, θα έπρεπε, που λέει ότι θα πρέπει να εξετάσουμε, να επανεξετάσουμε τις στρατιωτικές δαπάνες της Ελλάδας που είναι πάρα πολύ ψηλές και αν ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαμεσολαβούσε για την επίλυση των προβλημάτων με την Τουρκία και μεταξύ Τουρκία και Κύπρου, θα μπορούσαμε να εξοικονομήσουμε σημαντικό μερίδιο επί του ΑΕΠ, τουλάχιστον δύο ποσοστιαίε μονάδε επί του ΑΕΠ, και άρα θα βοηθούσαμε σημαντικά την Ελλάδα. Κυρία Στρέλα, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όσον αφορά το συμβούλιο αυτό. Εμένα οι προσδοκίες μου είναι πάρα πολύ χαμηλές γιατί υπάρχει ε, διαφωνία στην Ευρώπη. Αντί για το αποφασιστικότητα έχουμε δισταγμούς, αντί για αλληλεγγύη εγωισμούς και έτσι πορεύεται η Ευρώπη. Ας δούμε την ε, κατάσταση της Ελλάδας. Δεν θα μιλήσω για την Πορτογαλία, τη χώρα μου, γιατί μόλις ανέλαβε νέα κυβέρνηση. Οπότε το μόνο το οποίο μπορώ να κάνω να τους ευχηθώ καλή επιτυχία για το συμφέρον του πορτογαλικού λαού. Να αφαιρθώ λοιπόν στην Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν είναι μια τυχαία χώρα. Εδώ και δεκαετίες είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και του ευρώ και θα πρέπει να θυμόμαστε πως η Ευρώπη είναι βέβαια στο λίγνο της δημοκρατίας. Αυτοί οι παράγοντες ε, θα έπρεπε να υπαρκούν για να χαίρει σεβασμού από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Έλληνες ε, φέρουν ευθύνη για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται, αλλά το ίδιο ε, έχουν και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Ο κ. Φανδρέου έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να επιλύσει αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Ήταν θαραλέος, επέδειξε άξιο, πρέπεια, υιοθέτησε μέτρα λιτότητας που φτάνουν στα όρια του αδύνατου. Οπότε το ίδιο θα μπορούσε να συμβεί και στην Ιρλανδία ή και στην Πορτογαλία, στην Ισπανία ή στο Βέλγιο, στην Ιταλία ή στη Γαλλία. Οπότε ας ε, μου απαντήσουν το εξής ε, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Πώς θα μπορέσουν να δεχτούν τέτοια σκανδαλώδη επιτόκια αυτές οι χώρες και ταυτόχρονα να μειώσουν το χρέος και να αναπτυχθούν και να έχουν δουλειές οι χώρες αυτές ε, βρίσκονται σε δύσκολη θέση. Και τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Αν δεν τους σκοτώσει η αρρώστια θα τους σκοτώσει το φάρμακο. Οπότε χρειαζόμαστε ένα σχέδιο για να σταματήσει η κερδοσκοπία επί του κρατικού χρέους και να ξεμπροστιάσουμε τους οίκους αξιολόγησης. Ευχαριστώ. Κύριος Γκέρενς για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η πρώτη, το πρώτο προληπτικό μέτρο, όταν θέλει κανείς να αποφύγει μια μεγάλη πυρκαγιά, είναι να μην παίζει με τη φωτιά. Συμφωνώ με τον κύριο Μπαρός ότι θα πρέπει η ελληνική ε, κυβέρνηση να κάνει ό,τι μπορεί για να τακτοποιήσει τα του οίκου τη, έτσι ώστε και η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορεί να λάβει δράση με τη σειρά τη. Δηλαδή, με άλλα λόγια, η Ελλάδα πρέπει να ανακτήσει, να αποκαταστήσει την αξιοπιστία τη και απευθύνω έκκληση προς τους υπευθύνου, που αυτό σημαίνει προς όλους τους ηγέτες Ευρωπαϊκής Ένωσης και ρωτώ, έχουν συνέστηση των επιπτώσεων των δηλώσεών τους ε, ε, σε σχέση με την Ελλάδα τον, τον τελευταίο 18 μήνο. Πρέπει να σταματήσει πια αυτή ε, η, έκφραση διαφορετικών απόψεων και δηλώσεων αντιφατικών συχνά μεταξύ τους. Χρειάζονται λοιπόν τέσσερα πράγματα. Πρώτα ένα, ένα σχέδιο ουσιαστικό α, οικονομικής εξυγίανσης και ανόρθωσης, ευρωπαϊκή ε, ευρωζώνη και ευρωγκρουπ ενωμένο. Τρίτον, λίγο περισσότερο χρόνο από ό,τι αρχικά προβλεφθεί και τέτοια ιδιωτικοποίηση Και τέταρτον, αλληλεγγύη. Αλληλεγγύη καλώ νοούμενη. Που σημαίνει όχι μόνο νέα ε, οικονομική στήριξη, αλλά πάνω απ' όλα τεχνική στήριξη από πλευρά των εταίρων και δι τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Γκέρεν. Κύριο Ράγκελ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να πω το εξή. από το συγκεκριμένο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, δεδομένου και του κλίματος που βιώνουμε τις τελευταίες εβδομάδες, αναμένω μία απόφαση μεγάλης ευθύνης. Μεγαλύτερης ευθύνης από αυτή που αναλήφθηκε στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο ανέστηλε μόνο για λόγους εκλογικού χρονοδιαγράμματος μία απόφαση κατά τρεις μήνες. Θέλω να δώσουμε απόδειξη λοιπόν ευθύνη. Ε, τα οικονομικά και χρηματοπιστωτικά ζητήματα πρέπει να το αντιληφθούμε πλέον ότι αποτελούν ικανή και αναγκαία συνθήκη για το μέλλον τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά τα χρηματοπιστωτικό και οικονομικά ζητήματα είναι ένα μέσο για το βασικό στόχο τη Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι η διατήρηση τη ειρήνη. Εάν αντιμετωπίζαμε τα προβλήματα κατά τρόπον ώστε τα κράτη-μέλη να μην εμπιστεύονται αλλήλους δημιουργώντας και ε, εντείνοντας διαφορές μεταξύ των κρατών του Βορρά και του Νότου, των κρατών του Κέντρου και της Περιφέρειας. Θα οδηγήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση στην παρακμή της. Αυτό το οποίο διακυβεύεται στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο πέραν των τεχνικών ζητημάτων, πέραν ε, των ε, πολιτικών αποφάσεων, είναι να καθορίσουμε κατά πόσον θέλουμε το ευρωπαϊκό ε, οικοδόμημα να συνεχίσει να υφίσταται. Κατά πόσον είναι έγκυρο αυτό το ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τη διατήρηση της ειρήνης στην Ευρώπη. Αυτό είναι το θέμα. Εγώ διαπίστωσα σε πολλές ομιλίες των ηγετών είτε των χωρών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες είτε των χωρών που συνεισφέρουν ότι γίνονται ανεύθυνες ε, παρεμβάσεις οι οποίες πολλές φορές κάνουν έκκληση σε εθνικά και εθνικιστικά χαρακτηριστικά γεγονός που είναι πάρα πολύ αρνητικό. Κάνω έκκληση λοιπόν, μόνο αυτό να πω, ε, στην αίσθηση ευθύνη των Ευρωπαίων ηγετών, διότι θα πρέπει να βρουν λύσει οι οποίε θα οδηγήσουν την Ευρώπη στη διέξοδο από το πρόβλημα και σε μία λύση τη κατάσταση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πιτέλα για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Φόβος και αμοιβαία έλλειψη εμπιστοσύνη. Αυτό έλεγε προηγουμένω ο κύριο Μάουρου και αυτά είναι τα συναισθήματα που καθοδηγούν τι επιλογέ των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων για την κρίση. Νομίζω ότι η Ευρώπη μοιάζει με μια ομάδα ποδοσφαίρου που χάνει 2-0 και οι παίκτες της νομίζουν ότι μπορούν να γυρίσουν το παιχνίδι χωρί να κάνουν πάσε. Προσπαθώντα να βάλουν γκολ ο καθένα μόνο του. Μόνο του, κανένα δεν μπορεί να κερδίσει το παιχνίδι. Ακόμα και αν ήταν ο Μαραντένα και ο Πελέ εκεί να παίζουν, δεν θα μπορούσαν να κερδίσουν μόνοι του το παιχνίδι τη κρίση. Η ελληνική κρίση, καταρχήν, ήταν ε, διαχειρίσιμη. Εμείς όμως προχωρήσαμε και έχουμε φτάσει σε ένα πάρα πολύ δύσκολο σημείο και έχουμε, θα πρέπει να προχωρήσουμε βάζοντας στην άκρη επιζήμιες ζήλιες ε, και οικονομικές ε, απειλές. Πρέπει να το παραδεχτούμε. Πολλοί από του αρχηγού κρατών και κυβερνήσεων ε, αποδεικνύεται ότι είναι ηγέτες δεύτερη κατηγορία. Αντιμετωπίζουν την κρίση, λε, και είναι ευθύνη τη Ελλάδος. Δεν είναι ευθύνη των κρατών μελών και τη Ελλάδα. αλλά οικονομικών αγορών που μέχρι προχθέ δεν τι είχε ρυθμίσει κανεί. Τα κράτη, οι μέλη και οι ηγέτες μας ε, δίνουν και πάλι το δηλητηριασμένο μήλο και λένε ότι ή θα βελτιώσουμε τους δημόσιους λογαριασμούς και θα δούμε ποιος θα επιβιώσει. Δεν θα επιβιώσει κανείς και σίγουρα δεν θα επιβιώσει το ζωτικό κομμάτι της ευρωπαϊκής κοινωνίας. Χρειάζεται λοιπόν να στοχεύσουμε στην ανάπτυξη, να στοχεύσουμε ε, σε πόρους που θα οδηγήσουν στην ε, ε, έρευνα, στην κατάρτιση, στα μεγάλα δίκτυα. Και τέλος, για τη μετανάστευση, θα πρέπει να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν αγγίζει κανείς τη Σέγγεν το πολύ πολύ να την ενισχύσουμε. Την αφήνουμε όσο έχει, πρόκειται για μια σημαντικότατη κατάσταση, ε, κατάκτηση η οποία διατηρεί όρθια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει οι μεταναστευτικές ροές να διαχειρίζονται από την Ευρώπη μέσω μιας αρχής που θα περιλαμβάνει την ένταξη όλων, την ασφάλεια και την αλληλεγγύη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ Μαρινέσκου για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το Συμβούλιο περνά τις τελευταίες ημέρες της Ουγγρικής Προεδρίας και θα ήθελα να χαιρετήσω την ε, εύστοχη διαχείριση θεμάτων μερικές φορές καυτών από πλευράς της Ουγγρικής Προεδρίας. Θα δούμε αυτές τις μέρες τώρα εάν όντως επέτυχε ουσιαστικά αυτό το εξάμεινο, εάν δηλαδή τα κρατημέλη δεχθούν τις συστάσεις της Ουγγρικής Προεδρίας και αποδείξουν έτσι ότι είναι υπεύθυνα και στρατεύονται στο είναι εφαρμοσική του νέου μηχανισμού το πρόγραμμα ε, σταθεροποίησης και σύγκλησης, στα εθνικά προγράμματα είναι αναγκαία αλλά όχι επαρκή. Χρειάζεται συνένεση για την οικονομική διακυβέρνηση, κοινή οικονομική διακυβέρνηση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει καταβάλει σημαντικέ προσπάθειε και έχει καταλήξει σε μια συνένεση που πιστεύω θα εγκριθεί αύριο στην ψηφοφορία στην Ολομέλεια και ελπίζω το ίδιο πακέτο και το Συμβούλιο να το εγκρίνει, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερον, λόγος πολύ έγινε για, την, ε, για το χώρο Σέγγεν. Είναι πολύ σημαντικό ε, να αναγνωρίσουμε ότι χρειάζεται αναζωογόνηση αυτών των υφισταμένων μηχανισμών. Δεν χρειάζεται επανόρθωση των συνόρων μονομερής. Δεν αποτελεί αυτή λύση. Εάν ένα κράτος δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που, του, που έχει υπομειστεί στα εξωτερικά του σύνορα, θα πρέπει να του προσφέρουμε βοήθεια. Γι' αυτό άλλωστε υπάρχει και η Frontex. Αλλά δεν είναι δυνατόν να επανορθώνονται τα σύνορα. Και έτσι πρέπει το Συμβούλιο, με σύσταση τη Επιτροπής εφόσον χρειάζεται απολύτως να επιτρέψει με ενισχυμένη μας πλειοψηφία την επιστροφή ε, την επανόρθωση των σύνορων, αλλά όχι με μονομερείς λύσεις, γιατί αυτό δεν είναι λύση η μονομερής επιστροφή στα σύνορα. Η έκθεση της ε, Προεδρία ως προς τη στρατηγική ενσωμάτωση ε, υπέρ των Ρωμά και τα μέτρα για την εκείνη στρατηγική τη ζώνη του Δούναβη είναι πολύ σημαντικέ προτάσει. Για να προαχθούν όλε αυτέ οι πολύ σημαντικέ για την Ένωση προτάσει. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Ακολουθεί ο Κέλλαν. Ευχαριστώ. Κυρία Υπουργέ, κύριε Επιτροπή, η αδυναμία του Συμφώνου Σταθερότητας ήταν ένας παράγων της κρίσης αυτής, η οποία εξελίχθηκε και είναι πάρα πολύ σοβαρότερη. Κανείς δεν είναι αθώος ως προς αυτό. Έχουμε φτάσει τώρα σε μια κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, όπου η ελεγγύη και η ευθύνη είναι το μόνο που μετράει. Αλλά η αλληλεγγύη δεν σημαίνει ένα όλοι για έναν σημαίνει εξίσου και ένας για όλους. Κάθε κράτος μέλος πρέπει να λάβει ευθύνη για την ένωσή μας και να αρχίσει να δρά προς το κοινό καλό της Ευρώπης. Ναι, χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη και περισσότερη Ευρώπη σημαίνει περισσότερη πειθαρχία συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων μέτρων ε, κατά εκείνων που παραβιάζουν τους κανόνες. Για να αποκατασταθεί η αξιοπιστία της Ευρωζώνης, η Κομισιόν πρέπει να γίνει πιο ισχυρή και ανεξάρτητη για να μπορεί να ασκεί οικονομική καθοδήγηση και υποπτία. Η Κομισιόν έχει εντολή να αξιολογεί την κατάσταση στα κράτη-μέλη, να εκδίδει προειδοποιήσεις και συστάσεις. Αλλά το βασικό ζήτημα είναι η πολιτική βούληση και η ικανότητα να επιβάλλει πρόστιμα και αυτό θα πρέπει να γίνει κανόνας, όχι αντικείμενο πολιτικού παζαριού. Ο ρόλος του Συμβουλίου θα πρέπει ε, αντιστοίχως να μειωθεί σε διαδικασίες που οδηγούν σε κυρώσεις. Η αξιοπιστία της Ένωσης θα βελτιωθεί επίσης με την ποιότητα των στατιστικών, με το να αποκλείεται στο μέλλον οποιαδήποτε δυνατότητα παραποίησης τέτοιων δεδομένων. Η χώρα μου, η Εστονία, αντιμετώπισε βαθιά οικονομική κρίση πριν από τρία χρόνια. Όμως, εξορροπήσαμε τον προβλησμό και μπήκαμε στην Ευρωζώνη. Η Λετωνία επίσης ανέλαβε δράση και βρίσκεται σε καλό δρόμο. Όλοι για έναν και ένας για όλους. Όλοι πρέπει να μεταρρυθμίσουμε τις κοινωνίες μας. Να κόβουμε τις δαπάνες βεβαίως είναι οδυνηρό, αλλά είναι ο μόνος τρόπος για την ανάπτυξη και τη σταθερότητα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Κέλαμ. Περνάμε στη διαδικασία και τη Δίνω τον λόγο πρώτα απ' όλα στον κύριο Κέλλη. Ευχαριστώ και Πρόεδρε. Ακούσαμε σήμερα πάρα πολλά για το να δίνουμε, να δίνουμε, να δίνουμε και το να κόβουμε, να κόβουμε, να κόβουμε. Θέλω να προσθέσω μια άλλη διάσταση. Το ότι παίρνουμε και παίρνουμε και παίρνουμε. Και αναφέρομαι ειδικά στα επιτόκια τα οποία επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Τρική Τράπεζα στη χώρα μου, την Ιρλανδία, που προσπαθεί κάθε μήνα να επιτύχει τους στόχους της όσον αφορά τη, άδοση, τη διάσωση. Και αυτό δεν μας βοηθά. Ευτυχώς η Κομισιόν και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είδαν πως υπάρχει άδικη μεταχείριση. Τα επιτόκια αυτά αποτελούν μιλόπετρα στο λαιμό αυτού που πνίγεται, ενώ ταυτόχρονα στέλνουμε υποτίθεται τη σωστική λέμβο. Οπότε αύριο ζητώ από το Συμβούλιο να μειώσει τα επιτόκια της Ιρλανδίας και αν γίνει αυτό θα επιστρέψουμε στην ανάπτυξη και θα αποτελέσουμε ξανά μια χώρα περήφανη και μέλος της Ευρώπης. Σας ευχαριστώ. Τα Μπαϊντή. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρόκειται να υιοθετήσει τις προτεραιότητες της Ουκρικής Προεδρίας για την οικονομική διακυβέρνηση, για, τις, ε, για τη διαχείριση του προβλήματος στο Ρωμά και για την προσχώρηση της Κροατίας. Ο κύριος στόχος πάντως ήταν η έγκριση του πακέτου 6 νομοθετικών προτάσεων για την οικονομική διακυβέρνηση. Οι ειδικοί και διπλωματικοί της ε, Ουγγαρίας μπορούν να αισθάνονται πιστεύω υπερήφανοι γιατί έχουν ε, μπορέσει να διευθετήσουν πολλά από τα ζητήματα που έμεναν εκκρέμει μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου και έτσι μπορούν να προχωρήσουν ε, σε λύσεις συνενετικές στο δυνατό επίπεδο. Το ερώτημα είναι εάν η κυβέρνηση Ορμπάν έχει όμως αρκετή αξιοπιστία και πολιτική βαρύτητα ώστε να διαπραγματευτεί προτάσεις για το για την ολοκλήρωση αυτού του ευρωπαϊκού εξαμήνου και αν ο κύριος Μότο είναι εξίσου αξιόπιστος που είχε και την ευκαιρία νωρίτερα ελπίζω να τα καταφέρουν και οι δύο γιατί χρειαζόμαστε αυτό το πακέτο για την οικονομική διακυβέρνηση Ευχαριστώ τον κύριο Καταμπάιντε η κυρία Φιγκερή του έχει το λόγο Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε η κατάσταση είναι σοβαρή η οικονομική και η κοινωνική κατάσταση των περισσότερων κρατών μελών θα έπρεπε να ε, τύχει εξέταση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και να αναλυφθούν πολιτικές και κοινοτικές ευθύνες ε, για τα θέματα αυτά έχουμε μια πολιτική η οποία γίνεται όλο ένα και πιο φιλελεύθερη, ιδιωτικοποίηση ε, και νέε ανισότητε ε, και σε κοινωνικό, σε εργασιακό επίπεδο, περισσότερη ένδυα και κοινωνικό αποκλεισμό. Δυστυχώς, σε αντίθεση με τις μάχες που δίνονται και ε, τα όσα δίνουν οι εργαζόμενοι, ε, τι προτείνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να συνεχίσουμε με τις ίδιες νεοφιλελεύθερες πολιτικές που οδήγησαν σε κρίση την ε, Ελλάδα και την Ιρλανδία και απειλούν την Πορτογαλία και άλλες χώρες θα πρέπει να βρούμε άλλα μέτρα. Δεν θα πρέπει να ακολουθήσουμε τη συνήθη πορεία ε, νέων μέτρων που είναι χρήσιμα για το κεφάλαιο εις βάρος των εργαζομένων, των μικρογεωργών και των μικροεπιχειρηματιών που πλήττονται από αυτές τις πολιτικές λιτότητες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Και τώρα. Ε, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε η τωρινή πολιτική μεταναστευτική της Ένωσης είναι λανθασμένη όπως και αυτά τα οποία προτείνει η Κομισιόν περί εταιρικών σχέσεων για να δώσει μια νόμιμη χρειά στις μεταναστευτικές ροές από την ε, Βόρεια Αφρική. Επίσης αγνοούμε το ότι πάρα πολλές φορές έχουν να παλέψουν με μεγάλη ανεργία, ειδικά των νέων ε, ε, στη δε έχει διπλασιαστεί αυτή τα τελευταία 20 χρόνια. Οπότε αυξάνεται η πίεση δυστυχώς στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. Δεν χρειαζόμαστε περισσότερη μετανάστευση από τη Βόρεια Αφρική, αλλά στα μάτια της μετανάστευσης οι πολίτες μας δεν θέλουν τέτοια εταιρική σχέση κινητικότητας, αλλά εταιρική σχέση επαναπατρισμού. Θέλουμε σύνορα και ισχυρότερη Frontex. Frontex. Αυτό θα πρέπει να το εξετάσει η Σύνοδος ε, εκεί όπου συζητάνε τις λεγόμενες προόδους της μεταναστευτικής πολιτικής. Ευχαριστούμε κύριε Όμπερμαϊρ. Για ένα λεπτό η κυρία Κολάρας Καμπομπίνσκα. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ την περισσότερη ώρα μιλούσαμε για την ελληνική κρίση και δικαίως γιατί είναι τεράστιο το ζήτημα, αλλά ο πρόεδρος Μπαρόζο απίθυνε έκκληση και για στήριξη της ε, ζώνης Σέγγεν και βεβαίως ε, αυτό σημαίνει πως είναι πολύ δύσκολες συζητήσεις και δύσκολη η κατάσταση με τους αρχηγούς ε, κρατών. Οπότε για μένα που κατάγουμε από την Πολωνία και για τους Πολωνούς η ζώνη Σέγγεν και το ότι μπορεί κανείς να ταξιδεύει ελεύθερα στην Ευρώπη ήταν το σύμβολο της ελευθερίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μεγάλη κατάκτηση και πλεονέκτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ε, μπορούμε να δεχτούμε να περικοπεί γιατί ακριβώς ε, λόγω τέτοιων αποφάσεων βλέπουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση υπ' αυτό το Γι' αυτό λοιπόν ζητάω να υπερασπιστούμε την ε, ζώνη Σέγγιν και να συμπεριλάβουμε και τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία το συντομότερο δυνατόν. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Κολέσκα Βαβίτσκα. Κύριε Παπαδοπούλου, έχει το λόγο. Φέρτε ότι δεν είναι εδώ η κυρία Παπαδοπούλου. Ο κύριος Λιμπεράτσκι, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Στη διάρκεια της σημερινής συζήτησης, ε, με μεγάλη ικανοποίηση, διαπίστωσα ότι οι φιλελεύθεροι και οι αριστεροί άρχισαν να συζητούν το μέλλον της Ευρώπης και δεδομένων τα όσων ακούσαμε, ακούσαμε ότι η Ευρώπη απειλείται και θα πρέπει λοιπόν να αναλυφθεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα δράση. Φωνώ λοιπόν με τη δήλωση του κυρίου Μπαρόζο σήμερα ότι θα πρέπει να γίνει μια δήλωση σχετικά με το ε, φόρο για τις χρηματοπιστωτικές ε, συναλλαγές. Χαίρομαι που υπάρχει αυτό. Είναι κρίμα που δεν έχουμε ήδη ένα σχέδιο κειμένου. Αλλά τέλο πάντων το γεγονό ότι γίνεται ένα πρώτο βήμα είναι σημαντικό. Ε, πέραν τη Ευρωζώνη υπάρχουν και χώρε εκτό του ευρώ και θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν υπάρχουν προβλήματα και για τι συγκεκριμένε χώρε. Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ. Ο κύριο Κουμουτσάκο φαίνεται δεν είναι στην αίθουσα. Παρακαλώ. Ο κύριο Μπουσούτιλ να λάβει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για το θέμα της μετανάστευσης. Αύριο αναμένουμε ένα τριπλό αποτέλεσμα. Πρώτον, προστασία της ζώνης του Σέγγεν. Γιατί ισοδυναμεί με την ελευθερία για τους πολίτες του Σέγγεν. Είναι όντως ορατό το Σέγγεν για τον Ευρωπαίο πολίτη. Δεύτερον, περιμένουμε ευθύνε κοινέ υπευθυνότητα για τα εξωτερικά και όχι μόνο για τα εσωτερικά σύνορα και επίσης ζητούμε μια ισχυρότερη Frontex, περισσότερη λέγγυη και κοινή ευθύνη, διαμερισμό της ευθύνης. Όπως επίσης και περισσότερη συνεργασία με χώρες της άλλης όχθης της Μεσογείου, των, εκείνες τις χώρες δηλαδή που περούν μέσα από διαδικασίες επαναστάσεων. Αύριο λοιπόν για τη μετανάστευση χρειάζεται να επιδειχθεί πολιτική βούληση. Εάν λείψει αυτή, μπορεί να συνεχίσουμε να μιλάμε, αλλά δράση δεν θα αναλυφθεί. Ευχαριστώ κύριε Βουσούτιλ. Τέλος, να δώσω τον λόγο πρώτα απ' όλα στον επίτροπο τον κύριο Σαφκούτση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Νομίζω ότι η σημερινή ζωντανή συζήτηση αποτελεί απόδειξη ότι η μερίσια διάταξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι πολύ επίκαιρη και πολύ σημαντική για το μέλλον της Ευρώπης. Η Ελλάδα ήταν παρούσα στις περισσότερες παρεμβάσεις και νομίζω ότι η κατάσταση στην Ελλάδα είναι πολύ δύσκολη και δεν είναι εύκολες οι λύσεις. Συμφωνώ με όλους όσους είπαν όμως ότι είναι πολύ σημαντικό να αποδείξουμε στους Έλληνες ότι δεν έχουμε μόνο περικοπές και λιτότητα, αλλά υπάρχει φως στην άκρη του τούλερ και μπορούμε να βοηθήσουμε την Ελλάδα να επανέλθει στο δρόμο της ανάπτυξης. Η λιτότητα λοιπόν θα πρέπει να συνοδεύεται και από συγκεκριμένες πολιτικές και μέτρα και είμαι βέβαιος ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορούν να συνδράμουν την, Ελένα, την Ελλάδα, να αυξήσει τις δυνατότητές της, να απορροφήσει τα διαρθρωτικά ταμεία καλύτερα και να τα ε, εντάξει σε στρατηγικούς ε, τομείς υπέρ τη ανάπτυξη. Και μπορούμε να βοηθήσουμε τις ελληνικές αρχές να βελτιώσουν την ποιότητα τη συλλογή των φόρων. Ξέρουμε ότι μπορούμε να βοηθήσουμε τι χώρε να βελτιώσουν και το εκπαιδευτικό του σύστημα και μπορούμε να το κάνουμε αυτή τη στιγμή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι διατεθειμένη να προχωρήσει προ τη συγκεκριμένη άγουσα. Μπορούμε να ετοιμάσουμε προγράμματα τεχνική συνδρομή ε, που μπορεί να βοηθήσουν τα δύσκολα μέτρα λιτότητα που πρέπει να λάβουν οι ελληνικέ αρχέ. Και με αυτό θέλουμε να αποδείξουμε σαφώ ότι η Ευρώπη ενδιαφέρεται επιδεικνύει αλληλεγγύη και μπορεί να βοηθήσει όταν μια χώρα αντιμετωπίζει τόσες δυσκολίες. Νομίζω όμως ότι θα πρέπει να αποστείλουμε και το ίδιο μήνυμα ε, και να λάβουμε και το μήνυμα και από τις ελληνικές πολιτικές αρχές. Εμείς μπορούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, αλλά θα πρέπει και η Ελλάδα να επιδείξει ενότητα και να δείξει ότι είναι διατεθειμένη να αντιμετωπίσει τα δύσκολα ζητήματα που αντιμετωπίζει η χώρα και νομίζω ότι αυτή είναι η έκκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τους ε, εκπροσώπους ε, της Ελλάδος. Συνεργαστείτε, δείξτε μας την ενότητα και δείξτε μας ότι υπάρχει κοινή προσέγγιση σε αυτά τα τόσο ακαθόδη ζητήματα. Αυτή είναι η υπεύθυνη πράξη και έτσι θα πρέπει να προχωρήσετε. Πολλοί από εσά αναφέρθηκαν και στα πολύ ε, σημαντικά ζητήματα όπως είναι για παράδειγμα η λήξη του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Εδώ χρειαζόμαστε και τη βοήθεια των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα πρέπει να επιστρέψετε στι περιφερειά σα και να πείτε ότι έληξε το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και ξεκινάει ένα νέο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Διότι νομίζω ότι ξέρουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Υπάρχουν συγκεκριμένε συστάσει που απευθύνονται σε κάθε χώρα συγκεκριμένα, είναι πολύ ενδελεχής για κάθε χώρα, αλλά χρειάζεται πλέον η συνεργασία των εθνικών αρχών, των εθνικών κυβερνήσεων, προκειμένου να υπάρξουν αποτελέσματα και να γίνουν μεταρρυθμίσεις στα κράτη-μέλη. Μόνον έτσι θα μπορέσουμε να αλλάξουμε την ποιότητα και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας προς το καλύτερο και να ε, θέσουμε νέα όθηση στην ευρωπαϊκή οικονομία. Θα ήθελα να πω ότι για άλλη μια φορά θα προταθούν ε, ε, φόροι για τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. Πρέπει να γίνει μια πολύ διεξοδική αξιολόγηση αντικτύπου και αυτό νομίζω ότι θα είναι και μία από τις προτάσεις που θα κάνουμε, είναι και η συνεισφορά μας στην συνολική συζήτηση για αυτά τα τόσο σημαντικά ζητήματα. Η Ευρώπη θα έχει ηγετικό ρόλο και ελπίζουμε και ότι οι υπόλοιποι εταίροι μας διεθνώς θα μας ακολουθήσουν. Αρκετοί από εσά αναφερθήκατε στην περιοχή Σέγγεν και το γεγονό ότι πρέπει να υπάρχει ε, πολιτική υψηλή ποιότητα για τη μετανάστευση. Σας διαβεβαιώ ότι γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η ελευθερία και το δικαίωμα ελεύθερης μετακίνησης ε, στην Ευρώπη είναι ένα από τα πιο σημαντικά μας επιτάγματα και θέλουμε να το διαφυλάξουμε. Είμαστε διατεθειμένοι να το διαφυλάξουμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι θεματοφύλακα των συνθήκων και είναι διατεθειμένη να δράσει εάν αμφισβητηθούν τα προγράμματα αυτά. Από τις πρόσφατες εξελίξεις πρέπει να αναγνωρίσουμε επίσης ότι χρειαζόμαστε ε, συγκεκριμένες λύσεις για όλες τις πτυχές της μετανάστευσης και θα πρέπει να αποκαταστήσουμε και την εμπιστοσύνη στο σύστημα. Η, Ευρώπη είναι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγγνώμη, είναι πεπισμένη ότι μόνο μέσω συντονισμένης διαδικασίας ε, μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα παρά να έχουμε μονομερείς δράσει από πλευρά κρατών μελών για να επανέλθουν τα εσωτερικά σύνορα. Χρειαζόμαστε επίση μια πιο αποτελεσματική και πιο προστατευτική πολιτική και ελπίζουμε αυτό να λειτουργεί μέχρι το 2012. Αυτή είναι η πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ελπίζουμε να το υποστηρίξει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και τα κράτη-μέλη. Επιτρέψτε μου να πω και δύο λόγια για την οικονομική διακυβέρνηση και αυτό το νομοθετικό πακέτο των έξι προτάσεων, διότι ακούσατε κάποια πράγματα από τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα έχετε και την ευκαιρία να το συζητήσετε πιο αναλυτικά με τον συνάδελφο τον θα ήθελα να σταθώ σε ένα μόνο στοιχείο και αυτό είναι η σημασία του να υπάρχει συμφωνία το συντομότερο δυνατόν και όχι ε, καθυστερημένα, διότι ο χρόνος μας πιέζει και χρειαζόμαστε νέα μέσα για να οδηγήσουμε τις ευρωπαϊκές οικονομίες με καλύτερο και πιο αξιόπιστο τρόπο στο μέλλον. Μια καταλακτική παρατήρηση για την Κροατία. Νομίζω ότι θα πρέπει να συγχαρούμε την Κροατία διότι ε, οδεύει προς μια ιστορική στιγμή και νομίζω ότι αυτό θα αποτελέσει ένα πολύ θετικό μήνυμα όχι μόνο για όλους τους Κροάτες αλλά και για όλα τα Δυτικά Βαλκάνια. Θα ήθελα να συγχαρώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τον εισηγητή, τον κύριο Σβόμποντα αλλά και την Ουγγρική Προεδρία που έκανε εξαιρετική δουλειά και ε, προώθησε το συγκεκριμένο ζήτημα ώστε να καταλήξουμε και στα τόσο καλά αποτελέσματα ήδη από τώρα. Τέλος, να ευχαριστήσω την κυρία Ένικο Γκιόρη. Ε, πολλές φορές είπε ότι ήθελε να έχει μια προεδρία φιλική προς το Κοινοβούλιο και νομίζω ότι αυτό το απέδειξε με την τόσο συχνή παρουσία της εδώ και θα ήθελα να την ευχαριστήσω και με την για την εξαιρετική της συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Επίτροπε. Τώρα με το Συμβούλιο τον λόγο έχει η κυρία Γκιόρη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, Κύριε και κύριοι βουλευτές. Επειδή είναι η τελευταία φορά που μιλάω στην ε, Ολομέλεια, εξ ονόματος της ε, Προεδρίας, θα ήθελα να μιλήσω την ε, γλώσσα μου. Πολλοί είπαν πως η Ουγγρική Προεδρία έκανε καλή δουλειά. Σας ευχαριστώ για την αναγνώριση αυτή και τώρα γνωρίζω πως ε, πράγματι αξίζει κανείς να ε, σκεί μια προεδρία φιλική προς το Κοινοβούλιο. Ο κ. Μπαρός αναφέρθηκε στην εξάδα αυτή ε, το νομοθετικό πακέτο, ο κ. Σοκτρέπος αναφέρθηκε στην ένταξη Κροατίας και τους άλλους φακέλους, συναπόφαση όπως ξέρετε επιτρέπει στο Συμβούλιο και την Προεδρία να έρχεται σε επαφή με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να γνωρίζουμε τα θέματα που μας απασχολούν και αυτό είναι θετικό και για τις δύο πλευρές. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και για τη σημερινή συζήτηση όσον αφορά τις ε, θεμελιώδεις αξίες και αρχές ε, βλέπουμε μια συμφωνία, μια συνένεση. Είχαμε μια φιλοσοφική σχεδόν συζήτηση και χαίρομαι για το ότι έχουμε συμφωνία σε αυτά τα θέματα. Επίσης συμφωνούμε πως είναι πάρα πολύ δύσκολα ζητήματα αυτά τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσει το Συμβουλίο. Όσον αφορά το επίθετο ιστορικός, θα πρέπει να είμαστε πιο επιφυλακτικοί και φιδωλοί με την χρήση του. Συμφωνώ επίσης πως το πνεύμα του φόβου είναι κακό σύμβουλος οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης άρα θα πρέπει να το θυμούνται αυτό όταν θα συζητήσουν αυτά τα ζητήματα αύριο και μεθαύριο είναι πεποίθηση δική μου και της Προεδρίας πως πρέπει να οικονομήσουμε την ομιλία εμπιστοσύνη, την ευθύνη και την αλληλεγγύη. Αυτό πρέπει να κάνουμε ε, είτε μιλάμε για την οικονομική διακυβέρνηση, μεταρρύθμιση της ε, Σέγγεν, ε, σύστημα ασύλου ή την διεύρυνση. Πρέπει να βασιζόμαστε σε αυτές τις αξίες. Περισσότερη Ευρώπη, ισχυρότερη Ευρώπη, αυτό ζήτησαν οι περισσότεροι και το τελευταίο εξάμεινο σε αυτά βασιστήκαμε και εμείς Είμαστε πεπισμένοι πως η βαθύτερη ολοκλήρωση είναι η λύση στα προβλήματά μας. Τέλος, να αφερθώ στα ζητήματα τα οποία κληρονομήσαμε από τις προηγούμενες προεδρίες ως ε, Συμβούλιο. Έπρεπε να επιτύχουμε συμφωνία σε συγκεκριμένου φακέλους με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Να ξεκινήσω από τα οικονομικά. Μιλήσαμε ήδη για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Σεύτσοβιτς, τον κύριο Επίτροπο. Πράγματι, αξίζει να προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε στους πολίτες τι είναι το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Σημαίνει περισσότερη διαφάνεια, σημαίνει το να ξέρουμε τι κάνει το κάθε κράτος μέλος με τα οικονομικά του, με τον προϋπολογισμό του και είναι θετικό το ότι αφιέρωσε τόσο χρόνο στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυστηρότερη διαχείριση των προϋπολογισμών επίσης και η βάση ε, βεβαίως της ανάπτυξης βρίσκεται στην σκληρή δουλειά και την δημιουργικότητα. Να σας αναφέρω δύο λόγους ε, για τους οποίους θα πρότεινα να εγκριθεί η πρόταση αυτή που έχουμε μπροστά μας. Το είπα και το αυτό είναι καλύτερο από την αρχική πρόταση και σε όλα τα ζητήματα κάναμε παραχωρήσεις. στο Κοινοβούλιο. Ακόμα και στο θέμα της αντίστροφης ειδική πλειοψηφία κάναμε υποχωρήσεις. Ε, είπε ο κύριο Λάμσδορφ πως ε, ένα μόνο μέσο υπάρχει σε ολόκληρο αυτό το πακέτο και είναι αντίστροφη ειδική πλειοψηφία. Διαφωνώ. Το καλύτερο ε, χαρακτηριστικό αυτού του πακέτου είναι ότι υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας σε ολόκληρο το σύστημα που θα μας επιτρέψουν να αποφύγουμε κρίσεις όπως αυτή η οποία μας χτύπησε το 2008-2009 όσον αφορά την ελεύθερη μετακίνηση ανθρώπων. Να πω πως ε, στο Συμβούλιο Εσωτερικών στις 9 Ιουνίου καταφέραμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία για τα συμπεράσματα του Συμβουλίου η οποία διατηρεί την ε, ελευθερία αυτή γιατί έχουμε την δυνατότητα να προσαρμοστούμε στις νέες προκλήσεις και βεβαίως θα πρέπει να υιοθετούμε μέτρα εκτάκτου ανάγκης μόνο σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης και μόλις κατατεθεί μια πρόταση και αναμένουμε να γίνει αυτό το φθινόπωρο θα μπορέσουμε να δούμε τις λεπτομέρειές της. Μόλις με ειδοποίησαν πως παράλληλα με την ε, Ολομέλεια ε, το ανοιχτό ζήτημα που αφορούσε την ε, Frontex έχει επιληθεί οπότε σας ευχαριστώ για αυτήν την συνεργασία. Έκλεισε λοιπόν και το μόνο ζήτημα που είχε μείνει κρεμές. Το άλλο ζήτημα που είχαμε βέβαια ήταν να η δυνατότητα δανεισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας επιτύχαμε έναν συμβιβασμό με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έτσι θα μπορέσουμε να λύσουμε τα προβλήματα των χωρών της Βορειοαφρικής ε, μέσω ε, της, τράπεζας, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Αναφέρομαι σε αυτά τα οποία είπε ο κύριος ε, Ταμπαϊντή για τα κίνητρα τα οποία είναι εσωτερικά πολιτικά. Να ρωτήσει τους συναδέλφους του το τι ε, υπόθηκε στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων γιατί η ατμόσφαιρα εκεί ήταν τελείως διαφορετική χτες. Επίσης ο κύριος Ταμπαϊντή μπορεί να διαβάσει τις απαντήσεις των κρατών μελών στην ε, πρότασή μας. Μπορείτε να ασκήσετε κριτική βεβαίως σε αυτές τις ε, προτάσεις αυτό είναι το καλό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, το ότι συζητάμε τα πράγματα και συνεργαζόμαστε. Το άλλο το οποίο θα έλεγα στον κύριο Ταμπαϊντή είναι το εξής. Ένα από τα πιο θετικά σημεία της Ουγγρικής Προεδρίας, το κλειδί θα έλεγα της επιτυχίας μας, ήταν το ότι τηρούσαμε το πνεύμα των συνθήκων και σεβαστήκαμε τις αρμοδιότητες των διαφόρων θεσμικών οργάνων. Η εξάδα αυτή των μέτρων τώρα προχωράει και εμείς θα το παραδώσουμε στην επόμενη Προεδρία ξέροντας πως έχουμε κάνει ό,τι μπορούσαμε και ο κύριος Μπαρόζο και οι συνάδελφοι του επένεσαν την Προεδρία γι' αυτό και όλοι οι Ευρωβουλευτές επίσης στις επιτροπές. Ο κύριος Φαν ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, μπορεί τώρα να προχωρήσει όπως εκείνος ε, θεωρεί σωστό και τέλος. Να αφαιρθώ στην ένταξη της ε, Κροατίας. Ε, είπα πως πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και φιδωλοί με τη χρήση της λέξης ιστορικός. Αλλά στην περίπτωση αυτή πρόκειται για μια ιστορική στιγμή. Είναι σημαντικό αυτό μήνυμα για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων ότι έχουν δηλαδή μέλλον εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεθαύριο οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων ελπίζουμε να λάβουν την οριστική πολιτική απόφαση για την ένταξη της Κροατίας. Στις δε τελευταίες ώρες της Προεδρίας μας θα ολοκληρωθούν οι σχετικές συνομιλίες. Η Κομισιόν δουλεύει ε, όλο το 24ωρο έτσι ώστε η τελική έκθεση να είναι θετική, αυτή εκδόθηκε στις 10 ε, Ιουνίου και υπάρχει και μία ε, ομάδα εργασίας Συμβουλίου που συνεδριάζει κάθε μέρα για να ολοκληρωθεί αυτό το ζήτημα τέλος. Σας ευχαρίστησα ήδη, αλλά οφείλω να ευχαριστήσω και την Ισπανία και το Βέλγιο για την ε, συνεργασία στο πρόγραμμα του τρίου αυτού και εύχομαι κάθε επιτυχία στην Πολωνική Προεδρία που ακολουθεί. Ευχαριστώ κύριε Γκέρι. Ολοκληρώθηκε τη συζήτηση και περνούμε στο επόμενο θέμα της ημερησίας διάταξης. Πρόκειται για την έκθεση του συναδέλφου Ντέσσα, κοινή γεωργική πολιτική με χρονικό ορίστο το 2000.